Αγαπητοί συνάδελφοι, η μερίσια διάταξη είναι πολύ φορτωμένη. Γι' αυτό λέω να αρχίσουμε τις συζητήσεις μας τώρα. Το πρώτο σημείο προβλέπει την έγκριση. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν έξι τροποποιήσεις. Το εννέα για τις συμβιβαστικές τροπολογίες στην έκθεση Ντελή για την κοινωνική στέγαση. Θα το συζητήσουμε ως πέντε. Το δε έξι, ανταλλαγή από, απόψεων έκθεση Μορέν Σαρτιέ για την έκθεση ηλεκτρομαγνητικά παιδεία αναβάλλεται για αύριο και μετά το 17. Το 18. 18. Έκθεση ορί για τον προπολογισμό 14 και αυτό νωρίτερα. Το 13 έκθεση Χέντελ για τη διώσυνοριακές συλλογικές διαπραγματεύσεις αύριο το απόγευμα μετά την ψηφοφορία, δηλαδή μετά το σημείο 26 το 27 έκθεση τελή για την κοινωνική στέγαση κι άλλο. Θα είναι η πρώτη αυριανή ψηφοφορία του απογεύματο και το 28 ψηφοφορία για την έκθεση Κοστέλο Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων αναβάλλεται για την συνεδρίασή μας της 7ης Μαΐου. Τα υπόλοιπα θα κρατηθούν. Αν δεν υπάρξουν αν εγκρίνεται η απειλαγή αυτή. Ευχαριστώ. Και όσους μεταξύ προσήλθαν, λοιπόν, δύο, πέντε ανακοινώσεις. Πρώτον, έναρξη διαπραγματεύσεων για την έκθεση Σόγκορ για τα δημογραφικά στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη μετά από την απόφαση της Ολομέλειας την περασμένη Πέμπτη για την αναβολή της ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή Απασχόλησης θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο εν ώψη συμφωνίας με βάση την εντολή που έδωσε η Ολομέλεια. Και η διαπραγματευτική ομάδα θα αποτελείται από εμένα, και τον εισηγητή Σογκόρ, την κυρία Παπαδοπούλου για τους σοσιαλιστές, την κυρία Μάρκιν για τους φιλελεύθερους, την κυρία Ντελή για τους πράσινους, τον κύριο Τόμας Χέντελ για την ΚΟΕ. Ο πρώτος τριμερής διάλογος θα γίνει 13 Μαΐου 6 με 8 το βράδυ. Θα τα μάθετε βέβαια και όσο εξελίσσονται τα πράγματα. Δεύτερη ανακοίνωση. Η Επιτροπή μας θα εφαρμόσει τους νέους, τους νέους πώς να το πω έτσι, ε, νέους κανόνες διοργάνωσης των ήττα συνεδριάσεων. Ήδη έχουν πληροφορηθεί οι βουλευτές και εκλήθημεν να γίνουμε το πειραματόζωο των νέων αυτών μεθόδων για καλύτερη λέει πρόσβαση στα έγγραφα των συνεδριάσεων. Η εφαρμογή αυτή λέγεται e-meeting για να έχετε πρόσβαση σε φορητούς υπολογιστές και σε ταμπλέτας. Θα μπορείτε δε να κρατάτε τα έγγραφα αυτά για επόμενη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή αυτή παντού με Wi-Fi ή 3G, 3Z μάλλον. Η καινούργια λοιπόν αυτή η εφαρμογή υπάρχει ήδη από σήμερα, από αυτήν τη συνεδρίαση και μια ειδική πληροφόρηση θα διοργανωθεί εδώ μέσα αύριο για όσους το θέλουν μεταξύ 2 και 4 και 2 και 45. Ακόμα μαθαίνουμε λοιπόν σε μεταβατική περίοδο. Τρίτη ανακοίνωση. Όπως σας έχει ήδη δηλωθεί η γραμματεία της Επιτροπής μας και την ευχαριστώ γι' αυτό. Άρχισε να συντάσει ένα πληροφοριακό δελτίο όπως κάνουν και άλλες επιτροπές. Τέταρτη ανακοίνωση για τις ερμηνείες που ζητήθηκαν, διερμηνείες αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Για τους απόρους είχε ζητηθεί διερμηνία γαλλικά και αγγλικά στις 18 Απριλίου, άρχισε όμως μισή ώρα αργότερα από ό,τι προβλεπόταν με βάση απόφαση των σκιωδών της προηγούμενης. Άρα σπαταλήθηκαν ώρες διερμηνίας και επίσης μία διερμηνία γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά είχε ζητηθεί και ακυρώθηκε εκείνη η συνεδρίαση διότι δεν ήταν διαθέσιμη η Προεδρία. Πέμπτη ανακοίνωση. Γίνεται αναμετάδοση. Ο Λοιπόν, πάμε τώρα στο σημείο 3 και 4 που είναι κοινή συζήτηση των τροπολογιών των τροπολογιών για δύο κανονισμούς που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ε, κοινέ διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ταμεία μετά από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα ο κύριος Θωμάς Μάνης ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, στο θέμα δύο ανακοινώσει της Προέδρου έχω την εξής ερώτηση. Μόλις διαπιστώσαμε βάσει μιας έκθεσης ε, ποιοι συμμετέχουν στην Επιτροπολογία. Ε, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς. Ε, τώρα, τι γίνεται για τις χερσές μεταφορές η Επιτροπή Μεταφορών Μάλλον την εξυπηρέτηση εδάφους εννοεί ο μιλήτης. Εμείς κάναμε ένα συμβιβασμό με τεράστια ε, πλειοψηφία εγκρίθηκε κατά τρία τέταρτα, αλλά αυτό είναι μια εντολή για τη διαπραγμάτευση και ένα μήνυμα. Τι θα γίνει εκεί εάν ένας, ε, μία επιτροπή έχει προσφύγει στην παράγραφο 50, τι γίνεται στον τριμερή διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πρέπει να παρευρίσκεται. Κάποιοι μου είπαν από την Επιτροπή Μεταφορών ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό, θα το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να επαναστατήσουμε. Έχουμε μια κοινή απόφαση της Ολομέλειας με τεράστια πλειοψηφία. Μπορούμε να το απαντήσουμε τώρα, να το αναβάλουμε, δεν ξέρω, μια ερώτηση θέλω εγκαίρως να το θέσω ε, και στις ανακοινώσεις Προέδρου, γιατί ε, από κοινού καταφέραμε να επιτύχουμε αυτό το συμβιβασμό. Κοιτάξτε, δεν το ανέφερα αυτό καθόλου στις ανακοινώσεις μου, ξεχωριστό το ζήτημα το οποίο αναφέρεται. Κοιτάξτε, μπορώ να σας δώσω μια σαφή απάντηση εφόσον είμαστε η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για ένα μέρος του κειμένου αυτού το οποίο ενέκρινε η Ολομέλη, οποιοδήποτε και να είναι το αποτέλεσμα, εφόσον εγκρίθηκε η τροπολογία αυτή, ο εισηγητής από την Επιτροπή που είναι καθήλυνα αρμόδια προφανώς θα μπορεί να συμμετέχει στον τριμερή διάλογο. Είναι σαφές αυτό και προφανώς θα λάβουμε υπόψη μας τα αποτελέσματα αυτού του τριμερούς διαλόγου, κατά τη διάρκεια του οποίου ελπίζω ότι θα υποστηρίξουμε πραγματικά τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ ωραία. Περνάμε στο σημείο 3 και 4 της ημερήσιας διάταξης και, δώσ, και δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Τσαμπαορίμπα, ο οποίος ε, θα αντικαταστήσει και τον Αντάμ Κόζα και την Ελιζαμπέτ Μογάν Σαρτιέ και καθότι γίνεται κοινή συζήτηση θα δούμε πώς θα καταφέρουμε να διευθετήσουμε, να διαρθρώσουμε κάπως αυτόν τον διάλογο μονόλογο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όντως, όπως το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, εγώ αντικαθιστώ αυτή τη στιγμή τους δύο εισηγητές, η κυρία Ελιζαμπέτ Μογάν Σαχτιέ, και ο κύριος Αντάμ Κοζά με ενημέρωσαν για τις δύσκολες συζητήσεις στις οποίες συμμετείχανε, συζητήσεις και επαφές που είχαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κατάφεραν να καταλήξουν σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, τις οποίες σας προτείνουν να εγκρίνετε. Μία από αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες έχει να κάνει με την ηλικία την ηλικία η οποία αναφέρεται στο κείμενο, στο προτινόμενο κείμενο κανονισμού και στις δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για ένα όριο ηλικία το οποίο έχουμε στο κείμενο, κάτω από το οποίο οι νέοι άνεργοι μπορούν να υποφελούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Γίνανε διάφορες προτάσεις και επομένως η συμβαστική φυτροπολογία είναι πολύ σημαντική γιατί τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτό το όριο ηλικία, μάλλον χρησιμοποιούν πολλά διαφορετικά όρια ηλικία. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε μια συμβαστική πρόταση για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Επομένω, η συμβαστική πρόταση που κάνουμε εμεί είναι το όριο ηλικία είναι 30, 30 ε- έτη. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν θα πρέπει να απευθύνεται στους νέους κάτω των 30 ετών. Στη συνέχεια, θελήσαμε να δούμε ποιοι είναι οι τομείς δράσης για αυτή την πρωτοβουλία. Όντως υφίστανται κάποιοι ε, ορισμοί όσον αφορά τις περιφέρειες ΝΑΤΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θέλουμε να γνωρίζουμε αν στα πλαίσια μιας ε, περιφέρειας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πρωτοβουλία αυτή, αν δηλαδή μπορεί να αποφεληθεί κάποιο αυτή τη πρωτοβουλία και σε ποιο επίπεδο. Και προ αυτό γίνανε διάφορε προτάσει από του κοιόδη ηγητέ και η κυρία Μογάν Σαχτιέ και ο κύριο ε, Κόζα επέλεξαν την ακόλουθη λύση. Να προβλέπεται ένα ποσοστό της τάξης του 20%. Ως προς το 20% όμως αυτό, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι έχει γίνει και μία πρόταση από την ομάδα των σελιστών για να φτάσουμε το 22,5%. Και αυτό για τον εξής λόγο. Να μην λάβουμε μόνο υπόψη μας τις περιφέρειες αλλά και τις υποπεριφέρειες. Ως προς αυτό έχω κάποια ερωτήματα όσον αφορά τις υποπεριφέρειες δηλαδή. Ξέρετε ότι οι περιφέρειες ΝΑΤΣ έχουν σαφείς ορισμούς Ωστόσο, όσον αφορά τον ορισμό για τις υποπεριφέρειες, τα λεγόμενα sub-regions στα αγγλικά, εκεί υφίστανται ακόμα κάποιες αμφιβολίες και κάποια ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Επομένως, οι εισηγητές θα ήθελαν να γνωρίζουν ποιες είναι οι πρακτικές επιπτώσεις αν κάνουμε μια τέτοια αλλαγή. Δηλαδή, αν χρησιμοποιήσουμε την έννοια της υποπεριφέρειας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφύγουμε μία υποπεριφέρεια, για παράδειγμα πολύ μικρή με πέντε χωριά και μία κομμόπολη, με, με μια πολύ ψηλή ανεργία. Μάλλον στην περίπτωση αυτή θα πρέπει και αυτή η υποπεριφέρεια να μπορεί να αποφεληθεί από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Τώρα όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις. Όλοι συμφωνούσαν για τις προτινόμενες προϋποθέσεις. Τώρα, για την κατανομή των συγκεκριμένων κονδυλίων. Και γι' αυτό κάναμε μία πρόταση στα πλαίσια μιας επιστολής, την οποία απευθύναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία ζητάμε μία κατεπίγουσα διευθέτηση του ζητήματος αυτού προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε πρόσβαση στα απαραίτητα αυτά κονδύλια ήδη από την αρχή της περίοδου προγραμματισμού. Τώρα, όσον αφορά την απόρριψη της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας των μακροοικονομικών προϋποθέσεων, ομόφωνα απορρίψαμε την πρόταση αυτή. Οι τροπολογίες λοιπόν αναφέρονται σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία σας περιέγραψα και οι δύο εισηγητές, η κυρία Μογάν Σαχτιέ αλλά και ο κύριος Γκοζά, ζητούν μια ευνοϊκή υποστήριξη από την ε, Επιτροπή μας και ευελπιστούν ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Thank you very much. Just, just some, ε, Ευχαριστώ πολύ. Μερικά σχόλια μόνο επιπλέον η κυρία Γκιόνς. Ακόμα δεν έχει συμφωνήσει ε, το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο. Δεν είναι η συμφωνία αυτή, είναι η θέση του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή. Και είναι γεγονός ότι συμφωνήσαμε το ανώτατο όριο να είναι 30 για τους νέους και επίσης και για τους πτυχιούχους και για εκείνους που δεν έχουν άλλα προσόντα και δεξιότητες. Γιατί αυτό ήθελαν οι σκιώδεις ηγητές να συμπεριληφθούν. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία τα οποία προσθέθηκαν, ουσιαστική έγινε η συζήτηση. Από τη μια καταλήξαμε σε ένα συμβιβασμό λέγοντας ότι οι νέοι θα πρέπει να έχουν καλής ποιότητας μετεκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενδιάμεση δουλειά, όχι μια οποιαδήποτε προσφορά. Και επίσης η συμμετοχή τους δεν θα πρέπει να συνδέεται ή να είναι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε καταβολή άλλων επιδομάτων, είτε ανεργίας είτε άλλων κοινωνικών επιδομάτων και επίσης να δούμε να παίζει και ένα ρόλο το Κοινοβούλιο στην αξιολόγηση όλων αυτών. Δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα ενέχεται το Κοινοβούλιο, ακόμα το συζητάμε. Πάντως καταφέραμε να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και οι οργανώσεις νεολαίας και στι αξιολογήσει των προγραμμάτων αυτών. Αυτά πάνω κάτω για το συμβιβασμό. Ήθελαν όλοι πάρα πολύ να επιταχυνθεί η διαδικασία για να μπορέσει στις αρχές του 2014 να τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Um, thank uh, Ποιος θέλει το λόγο? Θέλω να μιλήσω κι εγώ, λέει η πρόεδρος. Άλλη, Σρότερ, άλλος, άλλος. Κλείνω τον κατάλογο ομιλητών. Ο Αλεχάνδρο Θέρκας και μετά η Ελίζα Σρότερ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Εξ ονόματος του Σέρχιο Γουτιέρες που πετάει και δεν μπόρεσε να φτάσει εγκαίρος, μου άφησε τις σημειώσεις για να πω για το θέμα αυτό. Υπάρχει πλήρη συμφωνία ε, την έκθεση Κόσα και τους συμβιβασμούς που έγιναν για τα διορθωτικά ταμεία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν θα πρέπει να αφήνουν απ' έξω ε, τους νέους 25 με 30 ετών που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, έβαλε και κριτήρια ποιοτικά, ε, αφαίρεσε ε, την επιφύλαξη ή το απόθεμα απόδοσης. Όλα αυτά τα, τα προγράμματα που προτείνουμε είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο ή μια εφετερία. Δεν είναι τερματισμός για να αξιοποιηθεί το κοινωνικό ταμείο. Και κάτι άλλο που θα μας απασχολήσει και σήμερα είναι ότι, όπως είπε και ο κύριος Τσαμπαόρη, θα πρέπει όσο γίνεται να διευρυνθεί αυτή η πρωτοβουλία και να καλύψει όσο γίνεται περισσότερες περιφέρειες. 22,5% είμαστε εμείς στην ανεργία αν κατάλαβα καλά το τι ζητάει το Συμβούλιο, ε, προτείνει 20%. Δεν έχουμε ακόμα τη μετάφραση στα ισπανικά, στα κείμενα. Τα 3 δις εκατομμύρια ευρώ που προβλέπονται για τους νέους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Είναι κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνο τον εισηγητή από ό,τι κατάλαβα για κοινή υποστήριξη από διάφορα ταμεία. Αλλά αν μειωθεί από μεταφερά πιστώσεων, αυτό το ποσό θα είναι πάρα πολύ μικρό τελικά. Επειδή υπάρχουν διάφορες εξαιρέσεις ήδη και μπορούμε να σας δώσουμε και τον κατάλογο των εξαιρέσεων, ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να φύγουν αυτά τα χρήματα και να πάνε ε, σε άλλα ταμεία από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ. Η Ελίζαπετ ε, Ευχαριστώ. Καταρχά ευχαριστώ πολύ όλους ε, τους εισηγητές του Σκιώδης. Κάναμε πολύ καλές διαπραγματεύσεις. Έτσι σε ηρεμία και νυφάλιε, προσπαθήσαμε πραγματικά να βρούμε την καλύτερη δυνατή διατύπωση. Ήταν πολύ καλό αυτό, πολύ σημαντικό. Το συζητήσαμε με την ησυχία μας και βγάλαμε καλού συμβιβασμού. Ιδιαίτερα όπω έχει τώρα η διατύπωση για την ηλικία, να το επαναλάβω, για να διαβεβαστεί στην εισηγήτρια μου φαίνεται πάρα πολύ καλή η παρούσα διατύπωση. Είναι καλή λύση και έτσι ε, θα πρέπει να εμείνουμε και απέναντι στο Συμβούλιο. Κάτι άλλο που κατά την άποψή μου δεν λειτουργεί, δεν αποδίδει, είναι ο συμβασμός ΔΕΛΤΑ, D, διότι εδώ γίνεται μία προσπάθεια, δεν εννοώ επί της ουσίας, συμφωνώ με την ουσία, αυτό που με προβληματίζει είναι το πρώτο τμήμα. Γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθεί το εθνικό με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν γίνεται για λόγους πρακτικούς. Έτσι όπως προτείνεται εδώ ΑΙ δεν λειτουργεί. Διότι αν κοιτάξουμε το άρθρο 100 ορίζει ε, την Επιτροπή Παρακολούθησης και Εποπτείας που είναι σε εθνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι και αντικείμενο διαπραγμάτευση αυτό στο ΣΥΠΙΑ και είναι και η επαναχώρηση σε σχέση με το κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχει μια μεγάλη εθνική και περιφερειακή συνεργασία, μετά λέει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν γίνεται αυτό, για λόγου πρακτικού. δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται. Λοιπόν, γι' αυτό είπαμε στι διαπραγματεύσει. θα το βάλουμε στο άρθρο 15, αλλά όχι στην πρώτη παράγραφο, αλλά στη δεύτερη και πέμπτη παράγραφο, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαρκώς να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα, να τηρείται ενήμερο, πας περιπτώσει, στην ετήσια έκθεση και στην έκθεση προόδου ε, και αλλάζουμε τη διατύπωση και λέμε ότι ενημερώνεται λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό λειτουργεί. Έτσι όπως το λέει τώρα η διατύπωση είναι ανέφικτο και εμείς οι πράσινοι δεν θα το υπερψηφίσουμε. Είχαμε βρει μια διατύπωση περί το τέλο των διαπραγματεύσεων να συμμετέχει πάντα το Κοινοβούλιο στι συζητήσει, αλλά δεν ήταν αυτό που, που έχει προταθεί τώρα. Αφήστε δε που δεν πρόκειται να περάσει από το Συμβούλιο. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η τεχνική δυνατότητα. Δεν υλοποιείται αυτό έτσι όπως προτείνεται εδώ. Να το ξανακοιτάξουμε παρακαλώ. Στην ίδια παράγραφο. Στην παράγραφο 2 και 5, στο ίδιο άρθρο δηλαδή. Και στην ετήσια έκθεση και στην έκθεση προόδου υποχρεωτικά να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο. Να έρχεται μια σύνοψη από κάθε περιφέρεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Και να αναθέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιφορτιστεί με αυτό. Μόνο έτσι ε, γίνεται η περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή συνεργασία. Μόνο έτσι μπορεί να συνδεθεί το ευρωπαϊκό επίπεδο με τα άλλα δύο. Παρακαλώ να το ξανακοιτάξουμε να ξαναβρούμε εκείνη τη διατύπωση που είχαμε βρει προς το τέλος των διαπραγματεύσεων για να το υποστηρίξουν και οι πράσινοι. Ιδιαίτερα το δεύτερο τμήμα το υποστηρίζουμε 100%. Αλλά αυτή η διατύπωση είναι κάτι το οποίο μας εκθέτει, διότι ζητάμε πράγματα που δεν προβλέπονται και δεν λειτουργούν. Bien, alors dans la vie, il faut... Λοιπόν, για να είμαστε συνεπείς, όπως η κυρία Σρέτερ, θα σας μιλήσω και εγώ για αυτά τα πράγματα. Αυτές οι ιστορίες με τις επιτροπές εποπτείας ή συνέχειας που δίνεται. Στις εκθέσεις Μορέν Σαρτιέ και Κόσα είχε πει τα ίδια πράγματα οι συνάδελφους. Εγώ δεν συμφωνώ όμως. Νομίζω ότι αυτά μπορεί να γίνουν σε κάποια άλλη ζωή, αλλά προς το παρόν διαφωνούμε. Οι επιτροπές αυτές Παρακολούθηση ή συνέχεια. Δέχομαι ότι έχουν κάποια χρησιμότητα, αλλά ο ρόλος των ευρωβουλευτών, όχι μόνο ω νομοθετών, αλλά και στις περιφέρειές τους, ότι πρέπει να παρατηρούν τουλάχιστον, να συμμετέχουν ως παρατηρητές σε αυτές τις επιτροπές, νομίζω είναι σωστό. Και το ίδιο ισχύει και για αυτή την περίπτωση που συζητάμε τώρα. Αλλά δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό, αλλά για δύο άλλα πράγματα. Πρώτον, ως μέλος της Επιτροπής μας και στο πνεύμα αυτό που είπε ο κύριος Σωρί η έννοια των υποπεριφερειών είναι κάτι που το θίξαμε και για την έκθεση της κυρίας Μωρέν Σαρτιέ για το Κοινωνικό Ταμείο, για τις περιαστικές περιοχές. Εγώ η περιφέρεια από την οποία εκλέγομαι, κανονικά δεν θα έπρεπε να εκλέγομαι. Γιατί αποτελεί ολόκληρο νομό που είναι ο φτωχότερος της Γαλλίας και άρα δεν έχει πολλές μεγάλες πόλεις και αυτό διότι το Ile de France όπως και σε όλη την Ευρώπη και τη Γαλλία είναι μέρος όπου συγκατοικούν οι πιο πλούσιοι με τους φτωχότερους. Δεν ισχύει αυτό μόνο για τον νομό Σεν Σεντενή, αλλά και για άλλους. Έχουν γίνει δύο φορές επισκέψεις του Αρμοδίου Επιτρόπου στο νομό αυτό Κουάνα Αγίου Διονυσίου στον Πομπινί και διαπίστωσε διεισόμασιν Γι' αυτόν τον λόγο ίσως δεν πρέπει να πούμε υποπεριφέρειες αλλά κάτι γενικά που να δείχνει ότι η κατανομή πρέπει, στις περιφέρειες πρέπει να ανταποκρίνεται κάπως στη διοικητική κατανομή που κάνουν τα κράτη. Vous souvenez que nous avions demandé que la commission emploi Τέλος, για να συνδεθούν αυτά που λέμε και με αυτά που συζητάει η Επιτροπή Περίφ, Ρέγγι δηλαδή. Να τα συνδέσουμε με κάτι που λέει σε ένα μία παράγραφο της έκθεσης Κόζα. Ο Επίτροπος λένε παραπονέθηκε και ζήτησε ότι πρέπει να συνδέεται και η δική μας επιτροπή και η δική μας επιτροπή λέγω ότι δηλαδή η περίφ πρέπει να λαμβάνει σοβαρά, να λάβει σοβαρά υπόψη της τη δική μας γνωμοδότηση και τα λέει τώρα και στα αγγλικά εδώ για να υπάρχει μια συνεπέστερη προσέγγιση η η Επιτροπή Περίφ πρέπει να ακολουθεί την Επιτροπή Απάσχα όσον αφορά το θέμα των διαθεσμικών συνεννοήσεων. Τελείωσε ο κατάλογος των ομιλητών, γι' αυτό τώρα θα ξαναμιλήσει ο κύριος Ορή. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατάλαβα πολύ καλά τα όσα είπε η Ελιζαμπέτ εξ ονόματος των Πρασίνων. Όντω. συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ε, συμβαστικές ε, προτάσεις των εισηγητών. Θα διαβιβάσω στους ε, εισηγητές όλες τις παρατηρήσεις σας και ελπίζω πραγματικά ότι θα καταφέρετε να υποστηρίξετε όλες αυτές τις προτάσεις που κάνουν οι δύο εισηγητές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τις δύο αυτές εκθάσεις, δηλαδή την έκθεση και την γνωμοδότηση αστικά, αύριο και θα καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε κατά αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα νέα στοιχεία στη διαπραγματεύσεις που θα κάνουμε με το Συμβούλιο. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. όπου θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης του κυρίου Ζόρς Μπάκα όσον αφορά την εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότηση, το οποίο θα υποβληθεί στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου η συγητή είναι ο κύριο Μαρινέσκου. Στο παρόν στάδιο θα εξετάσουμε τις 28 τροπολογίες που υπευλήθησαν, καθώς επίσης και τις τρει συμβαστικές τροπολογίες, τις οποίες υπέβαλε ο εισηγητής. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να επιμείνω στη σημασία αυτού του θέματος, ούτε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και συνδέονται με την εξωτερική πολιτική άλλων μεταφορών. Όπως είπατε, έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες, πολλές δικές μου από αυτές και από τη συνάδελφο Γιούτα Στάιμπρουκ ε, και τον κύριο Μπάνιον. Είναι 28 οι τροπολογίες τους ευχαριστώ όλους για την καλή συνεργασία μας. Από τις τροπολογίες καταφέραμε να καταλήξουμε σε τρεις συμβιβαστικές προτάσεις χωρίς ε, μεγάλες δυσκολίες, ακριβώς λόγω και της καλής μας συνεργασίας και χάρη σε αυτήν. Υπάρχουν κάποιες άλλες μεμονωμένες τροπολογίες που απομένουν και δεν καλύπτονται από το συμβιβασμό. Μπορούμε να τις υποστηρίξω ε, δεν βλέπω μεγάλες δυσκολίες γενικότερα, ούτε για την ψηφοφορία ε, που θα γίνει αύριο το απόγευμα. Με χαρά, αν έχετε ερωτήσεις, να τις απαντήσω. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή, λέει η κυρία Στένρουκ, και τον κύριο Μπάνιον. Πολύ καλά συνεργαστήκαμε όντως οι συμβιβαστικές τροπολογίες ήταν απαραίτητες. Αυτό που θέλαμε εμείς είναι οπωσδήποτε να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και οι κοινωνικοί εταίροι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η αγορά εργασία στην Ευρώπη και θα πρέπει να προσέξουμε. Το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα θέματα ε, με τις ε, υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους, το ground handling δηλαδή, και ε, για το ωράριο εργασία πληρωμάτων και κυβερνητών αεροσκαφών. Θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι μεγάλη η διεθνής ε, δραστηριότητα και ο ανταγωνισμός και δεν θα πρέπει να σηκώσει όλο το βάρο αυτού ε, ο κλάδο των εργαζομένων στι αερομεταφορέ. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που μπορούν να απαιτούν τα πληρώματα και οι κυβερνήτες. Και αυτό είναι θέμα δικό μας, της Επιτροπής μας, γιατί πρόκειται για θέματα υγιεινής και ασφάλεια στην εργασία και προστασία της υγείας των εργαζομένων. Και όταν έχουμε αερομεταφορείς από τρίτες χώρες που πετούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρούν ορισμένες προδιαγραφές, έτσι δεν είναι και συμβάσεις ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Αυτά. Κατά τα άλλα πιστεύω αύριο θα Πάνε όλα καλά στην ψηφοφορία, δεν έχουμε συγκρούσεις ε, και σταματώ εδώ. Ο κύριος Μπάνιο. Yes, uh, thank you. Um... Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Μπαχ και την Γιούτα Στάνμπρουκ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και όπως είπατε καταλήξαμε σε τρεις συμβαστικές προτάσεις οι τροπολογίε ουσιαστικά τόνισαν κυρίω το δυναμικό δημιουργία θέσεων απασχόληση στα πλαίσια του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού και επιπτώσει που θα μπορούσαν να είχαν και σε άλλου τομεί, βέβαια. Λέμε επίση ότι οι επενδύσει στι διασυνδέσεις των διαφόρων αεροδρομίων, ιδίω στι περιφέρειες εκείνες οι οποίε έχουν ανάγκη από περισσότερε επενδύσει, θα μπορέσουν να κάνουν τι περιφέρειες αυτέ λίγο πιο ανταγωνιστικέ και κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνει και μια καλύτερη κατανομή του πλούτου. Βλέπετε για παράδειγμα ότι στο Μένο Βασίλειο έχουμε το Λονδίνο, το οποίο είναι ένα κομβικό προφανώς αεροδρόμιο, ενώ απαιτείται μεγαλύτερη ανάπτυξη των περιφερειακών μας αεροδρομίων. Και ουσιαστικά αυτό θα αποφόρτιζε κάπως την ιδιαίτερη συμφόρηση που υπάρχει στο Λονδίνο και θα βοηθούσε οικονομικά και την περιφέρεια Βέβαια, έχω ακόμα κάποιε αμφιβολίε όσον αφορά την τροπολογία 19. Νομίζω ότι η Γιούτα πάντω θα ασχοληθεί περαιτέρω με αυτήν μέσω προφορική τροπολογία. Λέγεται ότι οι αερομεταφορεί θα πρέπει να συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαφόρων συμβάσεων. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να συνάδουν με τι συμβάσει αυτέ, εφόσον έχουν υπογράψει με αυτέ τι συμβάσει. Νομίζω πάντω ότι θα ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό λίγο αργότερα. Υπάρχει όμως μεγαλύτερο πρόβλημα με την τροπολογία 23. Λέγεται ότι οι αερομεταφορείς από τις τρεις χώρες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά προβλέπονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και πάλι όμως εξαρτάται από την τρίτη χώρα. Δηλαδή, αν είναι καταχωρημένες εκεί οι εταιρείε αυτές και αν η τρίτη αυτή χώρα έχει πραγματικά υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η εφαρμογή των ε, θεμελιωδών αυτών δικαιωμάτων εξαρτάται κάθε φορά από το αν το κράτος, το εν λόγω κράτος κάθε φορά έχει ε, υπογράψει την εν λόγω σύμβαση. Δεν ξέρω επίσης πώς θα μπορέσουν ποτέ να επιβληθούν κυρώσεις, ιδίως όταν μιλάμε για τρίτες χώρες. Αυτή είναι η διαπραγματευτική θέση την οποία έχουμε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε περισσότερο για τις διεθνείς αυτές ε, συμφωνίες αλλά βέβαια δεν μπορούμε εμείς να τις επιβάλλουμε. Δεν μπορούμε τουλάχιστον μέσω της ε, έκθεσης αυτής να καθορίσουμε το αν τρίτες χώρες θα απογράψουν όχι αυτές τις συμβάσεις. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλοι που θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Αν όχι, το, το λόγο έχει ο κύριος Μπακ Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μεγάλε δυσκολίε με αυτό. Θα πρέπει να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις να λαμβάνει υπόψη αυτά τα δικαιώματα και τα κράτη-μέλη να τα κατοχυρώνουν δεσμευτικά. Είναι πραγματικά θεμητό αυτό το αίτημα. Αν καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία και σε αυτή την νομοθεσία τελικά, ποιος είναι ο θεματοφυλάκας των συνθήκων, άρα και υπεύθυνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτά θα πρέπει να πείπτει και η αντίστοιχη ράβδος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε και την γνωμοδότηση αυτή αύριο και η Επιτροπή Μεταφορών θα ψηφίσει την έκθεση 7 Μαΐου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και όπως είπαμε στην αρχή της συνεδρίασής μας θα εξετάσουμε τώρα το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την 41 συμβαστικές τροπολογίες για την έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά την κοινωνική στέγαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει τις τροπολογίες αυτές, συμβαστικές τροπολογίες, στην συγγήτρια κυρία Καριμαντελή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το είπατε και εσείς ότι έχουμε 41 τροπολογίες. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές μου για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπένιον, τον κύριο Σέρκας, την κυρία Ζούμερ, Σόγκορα και την κυρία Μακάρθορ και θα ήθελα πραγματικά να πω ότι από την αρχή της εκπόνησης αυτής της έκθεσης, από τις πρώτες διαβουλεύσεις που είχαμε, πραγματικά καταφέραμε να κάνουμε μια πολύ καλή εργασία και συνεργαστήκαμε πολύ επικοδομητικά. Δυστυχώς, επί του παρόντος, δεν έχουμε λάβει ακόμα κάποια απάντηση από το ΕΛΚ για το 1 τρίτο του συμβιβασμού, ενώ η προθεσμία είναι σήμερα στις 4 το απόγευμα. Ακόμα λοιπόν και σήμερα δεν γνωρίζουμε για το 1 τρίτο τροπολογιών ποια είναι η τοποθέτηση, η οριστική θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Θα ήθελαν μη τι άλλο αύριο να υπερψηφίσουν το σύνολο των συμβαστικών τροπολογιών. Επίσης, για αύριο να ζητήσω από τους νησηγητές να απορρίψουν ε, τις τροπολογίε τροπολογίες εκείνες οι οποίες επιθυμούν την απόρριψη του κειμένου. Ξέρετε ότι το κείμενο αυτό, όπω σα είπα, αποτελεί την έκβαση μια πολύ συλλογική δουλειά ήδη από την αρχή τη όλη διαδικασία. Χρειαζόμαστε την έκθεση αυτή, γιατί το ζήτημα τη κοινωνική στέγαση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιρλανδία. Το ζήτημα τη στέγαση είναι πάρα πολύ σημαντικό, αποτελεί ένα αγαθό πρώτη ανάγκη και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει ένα ακόμα πιο δυνατό μήνυμα ότι η στέγαση αποτελεί θεμελιώδε δικαίωμα και η κοινωνική στέγαση μπορεί να μας βοηθήσει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την οικονομική, κοινωνική και οικολογική κρίση. Είναι πραγματικά μέσα από την κοινωνική στέγαση μπορούμε να δώσουμε μια ευρωπαϊκή λύση ακόμα και στο ζήτημα της ανεργίας. Η κοινωνική στέγαση αποτελεί απάντηση ακόμα και στο ζήτημα της απασχόλησης, της τοπικής απασχόλησης. Αξιοπρεπείς ε, θέσεις εργασίας οι οποίες θα βοηθήσουν προκειμένου να καταφέρουμε να βελτιώσουμε περισσότερο το οικονομικό περιβάλλον, για να δημιουργήσουμε επίσης πιο αξιοπρεπείς κατοικίε κατοικίες, με την απαραίτητη θερμική μόνωση, για παράδειγμα. Επίσης, η κοινωνική στέγαση αποστέλει ένα μήνυμα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Όντως, αγαπητοί συνάδελφοι, ο τομέας της οικοδομής αντιστοιχεί στο 40% των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε μέσω της κοινωνικής αυτής στέγασης να αντιμετωπίσουμε ακριβώς την αυτή πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή την ενεργειακή παινία που ε, ουσιαστικά αντιστοιχεί σε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε θέρμανση που δεν καταφέρουν να πληρώσουν τους ε, λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Επομένω, θα πρέπει αύριο να στείλουμε ένα μήνυμα προ Ευρωπαίου πολίτε, οι οποίοι πραγματικά μα έχουν ανάγκη. Μπορούμε να του στείλουμε αύριο ένα θετικό μήνυμα στα πλαίσια τη οικονομική αυτή κρίση που του αποσταθεροποιεί. Μπορούμε λοιπόν εμεί να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα ελπίδα και να πούμε ότι όντω η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σα βοηθήσει και μπορεί να σα δώσει συγκεκριμένε απαντήσει στην καθημερινή σα ζωή και να βελτιώσει το βιωτικό σα επίπεδο. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Σέρκα έχει το λόγο. Ναι, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω με ευχαριστίες για την κυρία Καρυματελή. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά της. 41 είναι οι συμβαστικές προτάσεις και χρειάστηκαν όλες αίμα, υδρότα και δάκρυα. Όλη αυτή η προσπάθεια οδηγεί σε μια σειρά συμβιβασμών όπου δέχεται όλες τις απόψεις με γενεοδορία Καμιά φορά χάνει την ε, συνοχή της η έκθεση από την πολύ γενναιοδορία και μεγαλοψυχία, γιατί τα έχει δεχτεί όλα η συγκητρία και ακόμα δεν ξέρουμε αν το ΕΛΚ συμφωνεί με τον τελικό συμβιβασμό. και τελικά κινδυνεύει η αξιοπιστία και η συνοχή της έκθεσης αν εγκριθούν ορισμένες συμβαστικές προτάσεις και χαθούν άλλες. Συμφωνώ και εγώ με την εισηγήτρια και απευθύνω έκκληση στο ΕΛΚ να δράξουν αυτή την ευκαιρία γιατί σε τέτοιους καιρούς κρίσης τόσοι Ευρωπαίοι άνδρες και γυναίκες υποφέρουν χάνουν το βασικό τους δικαίωμα ή αν δεν το χάνουν δεν είναι καν σε θέση να πετύχουν ένα αξιοπρεπές ε, ε, σπίτι ένα στοιχειώδη τρόπο στέγασης, θα πρέπει να προχωρήσουμε με προοδευτικό πνεύμα. Όπως είπε και η Καρίμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Τρεις είναι οι πραγματικότητες που συνδέονται μεταξύ τους. Η οικονομική κρίση, κυρίως σε πολλές από τις δικές μας χώρες, είναι το δράμα αυτό της ε, κερδοσκοπίας και της φούσκας στην οικοδομή. Καταστροφή. Έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς σπίτι και εκατομμύρια σπίτια χωρίς κατοίκους. Και μάλιστα τους πετάνε κάθε μέρα εξώσεις γίνονται. Ε, οι άνθρωποι που εργάζονται και δεν μπορούν να έχουν ε, ένα στοιχειώδες εισόδημα υπάρχει μια πραγματική αντίδραση, οργή λαού, γιατί το σύστημα εκτός του ότι είναι άδικο είναι και παράλογο από κάθε σκοπιά, από όπου και να το δεις. Είναι λοιπόν αυτό το οικονομικό φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο, αλλά και ένα τρίτο που είναι η κρίση ε, της κλιματικής αλλαγής. Αν έχουμε λογική πολιτική μπορούμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ για να μην χάνεται ενέργεια ή να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της ενεργειακής ε, παινίας τώρα στην κοινωνική στέγαση. Εμείς θα θέλαμε κάτι που έχει μπει λίγο στο συμβιβασμό, αλλά θα θέλαμε να τονίζει περισσότερο η έκθεση το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη στην κρίση αυτή και τις ευθύνες που φέρνει. Διότι δεν αρκεί, όπως κάνουμε καμιά φορά στις εκθέσεις μας, να λέμε διάφορες αιτιολογικές σκέψεις, λες και είμαστε πανεπιστήμιο. Κοινοβούλιο είμαστε εδώ πέρα. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, η παρατήρηση των προβλημάτων ω φαινόμενα. Θα πρέπει να προτείνουμε λύσεις, να δίνουμε λύσεις, όχι απλώς συστάσεις ή ευχολόγια ή γνώμες. Να λαμβάνουμε θέσεις στεναρές, ισχυρές. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να λαμβανουμε θεσεις στεναρε ισχυρε η τονίσει περισσότερο την ανάγκη μιας γνήσιας ευρωπαϊκής πολιτικής γιατί οι περιφερειακές δεν αρκούν. Δυστυχώς η Ευρώπη ε, για την κοινωνική στέγαση ε, έχει μια αλλοπρόσαλη πολιτική, για να μην πω ότι στερείται τελείως πολιτικής. Ε, έχουμε διαρθρωτικές πολιτικές, έχουμε κοινωνικές πολιτικές και πολιτική ανταγωνισμού πολύ σημαντική και αυτό εμποδίζει πολλά κράτη-μέλη, ακόμα και σε επίπεδο κράτους, να αναπτύξει μια ουσιαστική πολιτική κοινωνική στέγης σε κάποια τροπολογία θα ήθελα να μπει αυτό. Ε, δύο αρχές με κάθε σαφήνεια. Πρώτον, η Ευρώπη να μην είναι ο εχθρός και να μην εμποδίζει σε πολλά κράτη-μέλη. Έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική ανταγωνισμού που αντιτίθεται σε πολιτικές πολλών κρατών μελών και είναι παράλογη η θεώρηση για την κοινωνική στέγαση. Και δεν μπορούν να ε, ε, έχουν τα κράτη-μέλη μια κοινωνική στέγαση με κοινωνική ένταξη των πιο αποκλεισμένων. Ε, η πολιτική της Ένωσης οδηγεί σε γκέτο, σε εργατικές συνοικίες, σε εργατικές κατοικίες. Η κοινωνική στέγη είναι τελείως αποκομμένη από τα υπόλοιπα στρώματα του πληθυσμού. Τα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει παραπέρα, έχουν πιο ανεπτυγμένες πολιτικές τα λέμε έτσι έστω και χαλαρά και όχι με όσο σθένος θα θέλαμε, ε, το λέει πάντως ο συμβιβασμός να μην ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέματα επικουρικότητας. Και ένα τελευταίο, Πρόεδρε. Θα θέλαμε η Ευρώπη να έχει μια πολιτική που όχι απλώς να μην ενοχλεί, αλλά να βοηθάει ενεργητική. Γι' αυτό χρειαζόμαστε στρατηγική, συνοχή, παρατηρητήριο, ε, δεν προβλέπεται ε, στην έκθεση. Επίσης ζητούμε κονδύλια, αλλά να είναι και στην ημερήσια διάταξη, γιατί είναι εκατομμύρια Ευρωπαίοι, άνδρες και γυναίκες, που σήμερα δεν μπορούν να έχουν αυτό το στοιχειώδες δικαίωμα. Και όταν δεν έχει στέγη, πώς μπορείς να διεκδικήσεις άλλα δικαιώματα, υγεία, να δημιουργήσεις οικογένεια, να έχεις μέλλον και όραμα για τη ζωή σου, εν περιπτώσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, τελείως. Ah, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Τέλη για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι κάτι που το έχουμε υποστηρίξει εδώ και ε, τις τελευταίες εβδομάδες. τουλάχιστον την κύρια ιδέα όσο για τους συμβιβασμούς μπορούμε να υποστηρίξουμε πλήρως τους περισσότερους. Υπάρχουν και μερικά καινούργια στοιχεία βέβαια από τις συμβιβαστικές τροπολογίες που μας δυσκολεύουν. Ο εισηγητής ξέρει ότι η εισηγήτρια ότι ξέρει, ξέρει ότι δεν υποστηρίζουμε τους συμβιβασμούς HU και AM, τρεις από αυτούς. Και έχουμε μικρότερα προβλήματα με άλλους τέσσερις, με άλλες τέσσερις συμβιβαστικές του Δέλτα. Δεν μας ικανοποιεί η επίκριση που εκφράζεται εδώ των ε, μέτρων λιτότητας στη συμβιβαστική F η τελική φράση για την πολιτική ανταγωνισμού για τις δημόσιες υπηρεσίες επίσης μας δημιουργεί προβλήματα. Στο Ι, στον συμβιβαστική Γιώτα γίνεται μια παραπομπή με, στο σύμφωνο σταθερότητας που τη βρίσκουμε ανεπαρκή. Το υπόλοιπο του Γιώτα το δεχόμαστε αλλά για αυτό το τμήμα ακόμη το συζητάμε. Τέλος για τη συμβαστική σίγμα έχουμε αμφιβολίες ως προς τη, το νόημα της πρότασης κινητοποίηση των καταθέσεων. Τι ακριβώς εννοεί. Ίσως ε, είναι λίγο υπερβολική. Γενικά όμως 33 συμβιβαστικές τροπολογίες τις δεχόμαστε πλήρως. Τέσσερις περίπου και τρεις όπου έχουμε τεράστιες δυσκολίες. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά ακόμη μια φορά την Καρίμα και για τη συνεργασία της αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε γενικότερα γιατί ήταν πολύ προσινής προς τις τροπολογίες μας και προσπάθησε να συνεννοηθεί με τις περισσότερες ομάδες για να εγκριθούν όσο περισσότερες συμβαστικές γίνεται. Βέβαια πάντα υπάρχουν διαφωνίες πολιτικές για ορισμένα πράγματα γιατί είναι και τα προβλήματα δύσκολα. Πάντως έκανε μια πολύ καλή και τίμια προσπάθεια και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Η κυρία Γιαχούκα. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Και εγώ σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Είναι σημαντική και για άλλες επιτροπές. Και σε άλλες επιτροπές ζητούνται τα μέτρα λιτότητας και οι περικοπές. Η δική σας λοιπόν έκθεση είναι πολύ επίκαιρη. Η κοινωνική στέγαση φυσικά είναι βασικό στοιχείο για τη μείωση της ανέχειας των πτωχοτέρων. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που είμαι σε θέση να σας αναφέρω στο χάρτη της απορίας στην Ευρώπη της Ανέχειας που βρίσκονται οι πτωχότεροι και βρίσκονται έμαθα από μια αποστολή πολλοί στη χώρα μου σε μία από τις πλουσιότερες εισαγωγικά πόλεις ότι η κοινωνική στέγαση, το, τα αιτήματα για κοινωνική στέγαση έχουν αυξηθεί πάρα πολύ γιατί έχει αυξηθεί ανέχεια τα τελευταία χρόνια. Άρα είναι όντως επίκαιρη η έκθεση και έμαθα ότι τα τελευταία δύο χρόνια υπήρχαν μόνο δύο προσφορές διαμερισμάτων για μία πόλη 60.000 κατοίκων και με 43 υποψηφίους για το καθένα. Ελπίζω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα σας ακούσουν και θα χτίσουν περισσότερα κοινωνικά διαμερίσματα. Δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμη αντιστέκονται. Ευχαριστούμε. Μήπως το ΕΛΚ θα μας πει αν δέχεται τις συμβαστικές τροπολογίες ή ο Σκιώδης, ο Σκιώδης δηλαδή, ο Σκιώδης. Ο Σκιώδης. Ο κύριος Σογκόρν λείπει. Λείπει. Ο Ρή. Τέλο πάντων το θέμα ε, μήπως θέλετε να ξαναμιλήσετε κύριε Ωρή. Δεν ήθελα απλώς να πω ότι μέχρι τώρα ακόμη το συζητάμε, δεν έχουμε καταλήξει. Δεν συνεννοήθηκα ακόμη με τον κύριο Σογκόρν. Έχουμε μιλήσει αλλά δεν έχουμε ακόμη τελειώσει την ανταλλαγή απόψεών μας. Μέχρι αύριο το πρωί όμως θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Α, καλά. Σύμφωνα όμως με τους κανόνες που εγκρίναμε στους συντονιστές την περασμένη εβδομάδα, θα ξέρετε ότι η διορία μέσα στην οποία πρέπει να υποβληθούν οι συμβιβαστικές έχει λήξει και δεν μπορούν να αλλάξουν πια. μετά από τις τέσσερις την παραμονή της ψηφοφορίας. Ελπίζω λοιπόν ότι τελικά θα τα καταφέρετε λοιπόν η εισηγήτρια ξανά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βλέπω ότι όλοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα της κοινωνικής στέγασης και γι' αυτό καλώ και τους συναδέλφους του ΕΛΚΑ αύριο να καταφέρουν να εγκρίνουν πολλούς συμβιβασμούς, πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες γιατί για μένα ήταν πολύ δύσκολο να ικανοποιήσω τους πάντες λόγω έλλειψης χρόνου αλλά και δεδομένων και πληροφοριών και ακροάσεων και αλλά και η θέληση έλειπε μερικές φορές. Προσπάθησα να κάνω ό,τι έκανα ό,τι μπορούσα Ευχαριστώ και τους διοικητικούς υπαλλήλου και τους συνεργάτες μου χωρίς τους οποίους δεν θα είχα μπορέσει να κάνω τίποτα. Ευχαριστώ. Euh, Μάλιστα. Πολύ ωραία. Βλέπω λοιπόν ότι δεν είχατε τα απαραίτητα μέσα για να καταφέρετε να εκπονήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έκθεση αυτή. Είχατε βέβαια πάρα πολύ καλούς συνεργάτες από τη Γραμματεία και ξέρετε ότι ε, διοργανώσαμε και μία ακρόαση, καθώς επίσης και ανταλλαγή απόψεων, στο μέτρο του δυνατού βέβαια πάντα. Είμαι πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την έκθεση αυτή. Σε κάθε περίπτωση θα την ψεφίσουμε αύριο. και θα περάσει από την Ολομέλεια τον Ιούνιο. Περνάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Και είναι η σειρά μου να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο προφορικής ερώτησης, καθώς επίσης και ένα σχέδιο ψηφίσματος. Θα θυμάστε ότι ο Επίτροπος ήρθε για να μας παρουσιάσει μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά ένα σύμφωνο κοινωνικών επενδύσεων καθώς επίσης και τις κοινωνικές επενδύσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στα πλαίσια του συμφώνου αυτού. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στην ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Είπαμε αρχικά ότι θα μπορούσαμε να υποβάλουμε μια έκθεση πρωτοβουλία, Εν τέλει όμω αποφασίσαμε να εργαστούμε πιο γρήγορα, ακριβώ επειδή και η Ιρλανδική Προεδρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανακοίνωση αυτή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αποφασίσαμε να αντιδράσουμε μέσω προφορικής ερώτησης και μέσω ενός ψηφίσματο. Όσον αφορά τώρα την προφορική ερώτηση, θέτουμε ουσιαστικά τέσσερα επιμέρους ερωτήματα ερωτήματα τα οποία απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά, όπου ουσιαστικά θέλουμε να γνωρίζουμε πώς θα ενσωματωθεί αυτή η πρωτοβουλία για τις κοινωνικές επενδύσεις στις εργασίες εκείνες που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή για την ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Επίσης, θέλουμε να γνωρίζουμε πώς θα διαρθρωθεί αυτό το σύμφωνο κοινωνικών επενδύσεων με τους υφιστάμενους μηχανισμούς για την εφαρμογή της ε, στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020. Επίσης, ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς την πράξη θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτή τη στρατηγική για μια ενεργή κοινωνική ένταξη. Και τέλος, Απευθύνουμε ένα ακόμα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε φορά που αναφέρεται στα ομόλογα κοινωνικού αντικτύπου, στα ομόλογα κοινωνικών επενδύσεων, πώς θα μπορούσαν αυτά να εφαρμοστούν πάλι στην πράξη. Βάσει λοιπόν αυτών των προφορικών ερωτημάτων, θα κάνουμε μια συζήτηση και θα πρέπει να εγκρίνουμε και μια πρόταση ψηφίσματος, η οποία είναι αρκετά πλήρης γιατί απαρτίζεται από 55 παραγράφους και ουσιαστικά αναφέρεται σε μια γενική προσέγγιση για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια αναφέρεται σε επιμέρους σημεία στο ζήτημα της καταπολέμησης της ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα σημείο επί το οποίο η δική μας Επιτροπή έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία, το ζήτημα της καταπολέμησης της ειδική φτώχειας των παιδιών, αυτή που πλήττει δηλαδή τα παιδιά συγκεκριμένα και έπειτα μετά την έκθεση που μόλις τώρα εξετάσαμε, της ε, Καριμαντελή, αναφερόμαστε και στην έκθεση αυτή, στο ζήτημα, στο ζήτημα των αστέγων. Αναφερόμαστε επίσης στις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Αναφερόμαστε επίσης στη δέσμευσή μας για την υποστήριξη της απασχόλησης των νέων στην δυνατότητα της αγοράς εργασίας να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Αναφερόμαστε στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, στα ζητήματα που αφορούν τα δύο φύλλα. Επίσης, θέλουμε ένα ποσοστό 25% όσον αφορά την πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων και θέλουμε μια εκ των προτέρων χρηματοδότηση της εγγύησης για την ε, νεολαία. Τέλος, κάνουμε και κάποια αιτήματα όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Αυτές είναι οι βασικές κατευθυντήρες γραμμές του κειμένου αυτού, για το οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία τροποποίησης και έγκρισης για να καταφέρουμε να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Ουσιαστικά θέλουμε να παρουσιαστεί η έκθεση αυτή πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα ασχοληθεί με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και θα συνάδει κατά αυτόν τον τρόπο και με την πρωτοβουλία της Ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία, όπως σας είπα, υποστηρίζει ιδιαίτερα την πρόταση αυτή, την ακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω κάποιος συνάδελφος θα ήθελε να πάρει το λόγο, κύριο Στέρκας. Πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα να πω ότι η δική μου ομάδα φρονεί ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία αυτή που μας δίδεται ε, από τη συγκυρία και το χρονοδιάγραμμα το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού του Ιουνίου δεν έχουν πολλές ιδέες τώρα ε, για ε, τα κοινωνικά. Ο Βαν και η Σέρπα προετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη και μπορούμε ε, με την ανακοίνωση αυτή να ε, δράξουμε την ευκαιρία για να προτείνουμε κάποιες χρήσιμες ιδέες. Και γι' αυτό, κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ το χρονισμό μας. Δηλαδή, να μπορέσουμε να το εγκρίνουμε πριν τον Ιούνιο. Προσπαθούμε να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια για τον κοινωνικό πυλώνα της ε, ΟΝΕ και μάλλον αυτές οι δύο πρωτοβουλίες από κοινού θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να ακουστεί. Δηλαδή, αν δεν μιλήσει και το Κοινοβούλιο, αν δεν μιλήσουμε και εμεί, θα είναι μια κουφαντική εισηγή, η οποία θα είναι και σκανδαλώδη. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ. Εγώ μιλώ εξ ονόματος του Φίλιπ Ντεμπάκερ, ο οποίος ζητεί συγγνώμη για την απουσία του, αλλά είχε ε, μια υποχρέωση για τον τριμερή διάλογο της ΕΚΟΝ και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή μα συνεδρίαση. Ευχαριστεί το, την εισηγήτρια για το ψήφισμά τη. Ο κύριος Ντεμπάκερ πιστεύει ότι η καλύτερη προστασία από τη φτώχεια είναι το να έχει κανεί ένα δικό του σπίτι και ε, μια αξιοπρεπή δουλειά. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να υπάρχει παρουσία στην αγορά εργασίας ε, καλωσορίζει τις προτάσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ε, προαγωγή ε, και της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων αλλά και της επιχειρηματικότητας. Θα πρέπει να βοηθούνται όσοι βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση, αλλά να βεβαιωθούμε ότι το κόστος του συστήματος δεν διακυβεύει το σύστημα πρόνοιας για να μην στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κόστος εργασίας. Καλωσορίζει την πρόταση αυτή λοιπόν ο κύριος Δεμπάκερ και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξηθεί αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ε, των κοινωνικών πόρων. Οι κοινωνικές πολιτικές να μην υποστηρίζονται μόνο από το δημόσιο τομέα. Θα μπορούσε να υπάρξει καλή ε, ενεργή συνεργασία ΣΔΙΤ, δηλαδή ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ε, μέσω αυτών των δραστηριοτήτων. Θα κάνετε σχετικές τροπολογίες ο κύριος Ντεμπάκερ, αλλά επίσης πιστεύει ότι λίγε αλλαγέ πρέπει να γίνουν τονίζει, όπως έχουμε άλλωστε συζητήσει και στο παρελθόν, ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε οδηγία πλαίσιων για την ποιότητα και προσβασιμότητα ε, κοινωνικών υπηρεσιών ε, γενικού συμφέροντος. Τις επόμενες εβδομάδες θα επεξεργαστεί το θέμα. Αυτά λέγει ο κύριος Ντεμπάκερ και σας ανέγνωσα τα σχόλιά του. Να κάνω και ένα σύντομο σχόλιο δικό μου. Πιστεύω και ελπίζω να προχωρήσουμε προς ένα πακέτο κοινωνικών επενδύσεων που να μπορεί να συμπεριλαμβάνει και μέτρα για την ε, καταπολέμηση ε, της έλλειψης στέγης, του φαινομένου των αστέγων και ιδιαίτερα την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας ε, στα σπίτια για να μπορούν οι φτωχές οικογένειες, τα φτωχά νοικοκυριά να έχουν ε, μεγαλύτερο εισόδημα γιατί αυτή τη στιγμή δαπανούν πολύ μεγάλο εισόδημα ε, στην ενέργεια. Ελπίζω έτσι να τονώσουμε και τη ζήτηση στην οικονομία. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή αυτή. Άλλος κανείς θέλει το λόγο, Πρόεδρος, για αυτό το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων. Ποιος? ένα ράμπα του. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω την πρωτοβουλία αυτή. Πιστεύω ότι οι κοινωνικέ αυτέ επενδύσει είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικέ και η πολιτική που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή, η κοινωνική, δεν αποκρίνεται ε, στι προκλήσει τι οποίε έχουμε μπροστά μα. Όπω λέγεται στο σχέδιο ψηφίσματο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια αντικυκλική πολιτική να μην επηρεαστούμε από τις πολιτικές λιτότητες που δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο και να καταφέρουμε το κοινωνικό το ζήτημα να το θέσουμε στην καρδιά, στον πυρήνα πραγματικά των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζω λοιπόν πολύ στεναρά αυτή την πρόταση ψηφίσματος, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Κοστέλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω ελάχιστα πράγματα να πω, γιατί Ουσιαστικά έχετε καλύψει εσείς πραγματικά το μεγαλύτερο τμήμα της ανακοίνωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα ερωτήματα τα οποία τίθεται αυτή τη στιγμή θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερο και να αποσαφενίσετε κάποιες πτυχές της πρότασης αυτής. Λέγεται σε ένα σημείο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα δικό χάρτη για την ενεργή ένταξη. Δεν έχουμε συγκεκριμένε κατευθύνε γραμμέ. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι δείκτε για μια τέτοια στρατηγική ενεργού κοινωνική στέγαση. Ενδεχομένω όμω να πρέπει να επανεξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνεται πάντω μια τέτοια δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνεται ενδεχομένω μια κάποια εικασία στο δικό σα το ερώτημα. Ευχαριστώ. Euh, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι αναφέρεστε στην ερώτηση 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική διάσταση των εξειδικευμένων συστάσεων που γίνονται προς τα κράτη-μέλη. ιδίω όταν αυτά τα κράτη-μέλη υποβάλλουν εθνικό σχέδιο απασχόληση. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι τα εθνικά σχέδια απασχόληση που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη να έχουν και μια έντονη κοινωνική διάσταση. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένει να υπάρχει μια καλύτερη εξισορρόπηση του μείγματο πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και επιμένουμε και στο ζήτημα αυτό, στις σχέσεις που έχουμε και στις επαφές που έχουμε με τα εθνικά κοινοβούλια. Θα εξετάσουμε πάντως περισσότερο τις τροπολογίες σχετικές, οι οποίες θα υποβληθούν μέχρι τις 26 Απριλίου. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και μόνο στα αγγλικά μπορούν να υποβληθούν οι τροπολογίες αυτές, τις οποίες στη συνέχεια θα εξετάσουμε. Όσον αφορά την προφορική ερώτηση, θα εξετάσουμε τις σχετικές τροπολογίες στις 7 Μαΐου και θα τις εγκρίνουμε αμέσως, προκειμένου να καταφέρουμε να πάμε στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Και όσον αφορά τις ε, τροπολογίες για το σχέδιο ψηφίσματος, θα εξετάσουμε σε 7 Μαΐου τις ε, σχετικές τροπολογίες, αλλά μέχρι τις 29 και 30 Μαΐου θα έχουμε διορία για να τις ψηφίσουμε και για να εγκρίνουμε κατά αυτόν τον τρόπο το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος και που θα συνοδεύεται από το προφορικό ερώτημα το οποίο σας ε, παρουσίασα. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Και περνάμε τώρα στο σημείο 8, στο οποίο θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την συνάδελφό μας από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, την κυρία Αν Γένσεν, γιατί καλώ ήρθατε καταρχάς αγαπητέ συνάδελφοι, είστε η Γενική Συγγήτρια του Σχεδίου Προϋπολογισμού για την, το, το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014 Είστε λοιπόν η Γενική Εισηγήτρια Αρμόδια για το Σχέδιο Προπολογισμού 2014 και συνεργάστε μαζί σας ο κύριος Όρη. Θα σας δώσω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο για να μας πείτε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, καθότι γίνανε αλλεπάλληλες συζητήσεις για τον προπολογισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς λοιπόν θα έχει ο προπολογισμός το 2014. Έχετε το λόγο. Ε, yes, ε, Σας ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε έναν θετικό προπολογισμό για το 2014. Ψηφίσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές στην Ολομέλεια του Μαρτίου, όπου είπαμε ξεκάθαρα ότι ξεκινάμε με πάρα πολλές δυσκολίες. Και αυτό γιατί δεν έχουμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι σχετικές συζητήσεις με το ζόρ έχουν ξεκινήσει. Δεν έχουμε νομική βάση επίσης για τις γραμμές του προπολογισμού. Και θα πρέπει να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τα 70 περίπου διαφορετικά νομοθετικά κείμενα τα οποία έχουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μέσα σε όλες αυτές τις δυσχέρειες πρέπει να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για τον ετήσιο προπολογισμό για το 2014 και έχουμε και αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν έχει επιληθεί όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεκινήσει το έτος 2014 με πάρα πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι δεν θα έχουν πληρωθεί ήδη από το 2013 ακόμα και παλαιότερους. Και γι' αυτό τον λόγο καταλαβαίνετε ότι εκκρεμούν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν και τα οποία σχετίζονται με τον ετήσιο προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία ενδεικτική κατάτμιση του προπολογισμού από τα κράτη-μέλη όσον αφορά το πολιετές πλαίσιο. Και εκεί πέρα μπορεί να δει κανείς αν τελικά οι προτάσεις αυτές συνάδουν με τα δικά σας συμφέροντα και τους δικούς σας τους στόχους, αυτούς που προωθείτε κι εσείς ως Επιτροπή για κάποια προγράμματα, προφανώς για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και για πολλά άλλα προγράμματα στον κοινωνικό τομέα. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν ίδια εισηγήτρια προπολογισμού για την Επιτροπή αυτή, επομένω έχω παρακολουθήσει εκ του σύνεγγις κάποια από τα προγράμματα αυτά τα οποία, με τα οποία εσείς ασχολείστε και προφανώς τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν και στο μέλλον. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς μια ξεκάθαρη εικόνα του πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω ότι προχωράμε μπροστά χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πού πηγαίνουμε. Είμαι πάντως εδώ για να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για τα τμήματα του προπολογισμού που σας αφορούν. Θα ήθελα να σας δώσω και κάποιες πρακτικές πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για τον προπολογισμό του 2014, κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη Μαΐου. Αυτό μας έχουν πει ενδεικτικά μέχρι στιγμής και εμείς προτείναμε να χρησιμοποιήσουν την πρότασή τους για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ως σημείο εκκίνησης για τον προπολογισμό. Και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι ε, έχουν συναντηθεί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και έχουν λάβει κάποιες απόψεις τι οποίες ενδεχομένως να λάβουν υπόψη του ή να τις συμπεριλάβουν στην πρότασή τους. Δεν ξέρουμε όμως αν οι ε, στόχοι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο σας έχετε προωθήσει πάρα πολύ ως επιτροπή, αν θα ευοδοθούν οι στόχοι αυτοί. Και ξέρω ότι εσείς ε, διαπραγματεύεστε μέσω των νομοθετικών κειμένων το ζήτημα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Μέχρι τα τέλη πάντως Μαΐου θα έχουμε μία πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, το αργότερο το Μάιο θα πρέπει να υποβάλλετε εσείς κάποιες ε, ιδέες ή προτάσεις όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, τις προπαρασκευαστικές δράσεις, γιατί ακόμα ελπίζουμε ότι θα υπάρχει δυνατότητα να αναλύσουμε κάποιες νέες ιδέες ακόμα και στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, τουλάχιστον αυτό θα προωθήσουμε εμείς σαν στάση. Γι' αυτό γιατί θα πρέπει να υποβληθούν και αυτές οι προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τοποθετηθεί στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις αυτές. Ξέρετε ότι θα πρέπει απλώς να υποβάλλετε μία σύντομη πρόταση όπου θα λέτε ποια πιλωτικά προγράμματα, η ποιες προπαραβασκευαστικές δράσεις θέλετε να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας πει αν είναι δυνατόν να προωθηθούν τα προγράμματα αυτά, αν ήδη καλύπτονται από κάποια εφιστάμενα προγράμματα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που έχουμε επιτάπητος, επί του παρόντος. Θα ακούσω πάντως τώρα την παρέμβαση του κυρίου Όρη και τους υπόλοιπους συναντέλφους στη συνέχεια και θα επανέλθω βέβαια στο ζήτημα αυτό και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της όλης διαδικασίας, ευελπιστώντας ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία. Έχουμε φτάσει πια στο σημείο αυτό που έχουμε πια μια πάρα, μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Προπολογισμών και των Εξειδικευμένων Επιτροπών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη διαδικασία εκπόνηση του προπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σωρή και μετά ο Φρεντέρικ Νταχτέν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την κυρία Γένσεν για τις πληροφορίες που μας έδωσε και την ενημέρωση. Συμφωνώ απολύτως ότι η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη όσο και λεπτή. Διότι είναι λίγα τα στοιχεία που έχουμε και πληροφορίες ε, με βεβαιότητα. Ακόμα και κάποια στοιχεία που φέρνονται δεδομένα και βέβαια στη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου είναι στον αέρα. Γίνεται λόγος για μια ρήτρα ευελιξίας. Τι στο καλό είναι αυτό το πράγμα στον προϋπολογισμό του 2014 αν υπάρχει ρήτρα ευελιξίας, θα επηρεάσει ακριβώς τη σχέση που έχει ο προϋπολογισμός του 2014 με ε, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα υπάρξει ενδεχομένως ένα περιθώριο χειρισμών ή ελιγμών μεγαλύτερο. θα δείξει ε, που θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε τώρα είναι ένα κατάλογο προτεραιοτήτων. Τι θέλουμε εμείς να δούμε στον προπολογισμό του 2014 να συμπεριλαμβάνεται. Η Επιτροπή Απασχόλησης δεν είναι βέβαια η μόνη επιτροπή που θεωρεί ότι για την επόμενη προγραμματική περίοδο ή και για τον επόμενο προϋπολογισμό το κλειδί είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας η αύξηση της ευημερία και της ανάπτυξης όχι μόνο χάρη στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020 αλλά για το μέλλον της Ευρώπης αυτό που έχει σημασία είναι η ανάπτυξη ε, η μεγέθυνση της οικονομίας. Αυτό είναι το κλειδί και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε και όλες τις πρωτοβουλίες που δημιουργούν εργασία. Θέλουμε όμως και αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τα διαστατικά ταμεία και να χρησιμοποιούμε με τρόπο πιο στοχευμένο τα ταμεία αυτά για να προωθούμε την ανάπτυξη. Αλλιώς δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας χωρίς οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς σήμερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζωφερή. Αυτό που θα θέλαμε εμείς να δούμε να ε, ε, δημιουργούνται προγράμματα ενεργούς ενίσχυσης απασχόλησης. Επίσης θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανέργους ε, για να μπορούν να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι άνεργοι είναι όλο και πιο μακροχρόνιοι άνεργοι παραμένουν σε ανεργία και όσο περισσότερο χρόνο είναι εκτός αγοράς, ε, τόσο πιο δύσκολο είναι να επανέλθουν και ψυχικά και ως προς το ηθικό τους, αλλά και οι γνώσεις τους ε, καθίστανται απαρχιωμένες και δεν μπορούν στη συνέχεια να μπουν σε μια εξελισσόμενη ε, αγορά εργασίας. Και εκεί χρειάζονται βοήθεια στην επανένταξή τους, στην επιστροφή στην απασχόληση και στην ενεργό εργασία. Ξέρω ότι προετοιμάζεται αυτό το καιρό ε, μια μεταρρύθμιση και του Eurest για την πρώτη θέση εργασίας, για την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες για την νεολαία και για να βρίσκουν δουλειά οι νέοι και αξίζει να τις υποστηρίξουμε και όλες τις δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Πέρα από την απασχόληση και την ανάπτυξη πρέπει να βελτιωθούν και οι δυνατότητες απασχολησιμότητας λεγόμενης γιατί εκεί υπάρχουν όλο και περισσότερο Δηλαδή, πολλοί είναι εκείνοι που ψάχνουν δουλειά, αλλά δεν βρίσκουν δουλειά γιατί δεν έχουν τι απαραίτητε δεξιότητες και προσόντα. Γιατί υπάρχουν εργοδότες που ψάχνουν εργαζομένους και δεν βρίσκουν κόσμο να καλύψει τις θέσεις εργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν και πάλι στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση. Εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε και στον προϋπολογισμό του 2014 αυτό που χρειαζόμαστε είναι πιστώσεις. Πέρα από όλα αυτά, πρέπει να στείλουμε και ένα συμβολικό μήνυμα, που δεν είναι μόνο συμβολικό, είναι και ουσιαστικό. Και έχει και πραγματική χρησιμότητα. Δηλαδή, έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Κάποια στιγμή ακούστηκε ότι αυτό θα καταργηθεί. Εμείς θέλουμε να έχει αρκετές πιστώσεις πληρωμών, να διατηρηθεί βέβαια αυτό το ταμείο ε, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και να θυμίσω ότι επί σειρά ετών ακούγαμε επικρίσεις ότι εντάξει αυτό το ταμείο είναι μείον αλλά και αυτά τα λίγα κονδύλια που έχει υποπορροφούνται. Μπορεί αυτό να συνέβαινε στο παρελθόν. Σήμερα δεν ισχύει. υπάρχουν όλο και περισσότερες ανάγκες και όλο και περισσότερες αιτήσει για ε, να επιφοηληθεί κανείς από το ταμείο αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να παραμείνει η απαραίτητη αυτή η αντίστοιχη γραμμή στον προπολογισμό του για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Επίσης, η ανάληψη υποχρεώσεων και οι πληρωμές θα πρέπει να διατηρηθούν ε, ε, ιδιαίτερα για τη βοήθεια που χορηγεί η Ευρώπη στους απόρους και στους πιο ευάλωτους. Ακόμα δεν έχει εγκριθεί αυτή η έκθεση, επίκειται, τον επόμενο καιρό θα εγκριθεί. Σήμερα η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποστηρίζει εθελούσια συμμετοχή ε, σε αυτό το ταμείο για τη βοήθεια προς τους πιο ευάλωτους. Πρέπει να βρούμε μια λύση, την κατάλληλη λύση, που να μπορούν να δέχονται και τα κράτη-μέλη και να την υποστηρίξουν για να έχει και τους απαραίτητους πόρους ε, για να ανταποκρίνεται στην αποστολή. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Προς το παρόν δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε λύση για αυτό το συγκεκριμένο ταμείο. Οι διάφορες έχουν στείλει τις σκέψεις τους και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να έχουμε καταλήξει. Επί σειρά ετών, από την πρώτη μου θητεία θυμάμαι εγώ, αλλά και στην προηγούμενη θητεία, συζητούσαμε συνέχεια για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής ΙΜΚΟ για την προώθηση και προαγωγή των μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων, για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων. Όλες αυτές είναι επιχειρήσεις που δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Και οι πολύ μικρές και οι λεγόμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, οι καινοτόμες Όλες αυτές θέλουν και αξίζουν υποστήριξης και ενίσχυση. Αυτή η ενίσχυση θα πρέπει να προέρθει από τον προϋπολογισμό του 2014. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Διότι <laughs> όλα αυτά ανήκουν στις εξουσίες και στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Θα πρέπει να βοηθήσουμε, να πιέσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να οδεύσουν όλα προς την ίδια κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεν αρμοδιότητες αλλού, ας πούμε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, την υγεία των εργαζομένων και εκεί οφείλει το Κοινοβούλιο να παρεμβαίνει. Για να έχουμε τους απαραίτητους πόρους έτσι ώστε να ε, προάγουμε την προστασία των εργαζομένων. Και δεν θα πρέπει όταν λήξει αυτή η κρίση να έχουμε πιο επισφαλείς θέσεις εργασίας για τους εργαζομένους από ό,τι πριν την κρίση. Αυτά ήθελα να σας πω, αυτά επιθυμώ να δώσω στον προπολογισμό του 2014. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων αυτή που έχουμε, αλλά από ό,τι βλέπω η Επιτροπή Απασχόλησης συμφωνεί πάνω κάτω με τις ιδέες της ηγήτρας. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στο Φρεντερίκ Νταρντέν. Πρώτα όμως να πω στην κυρία Γένσεν ότι όσον αφορά το Ταμείο για τους Απόρους, τους πιο ευάλωτους, η θέση του κυρίου Ορή είναι θέση του κυρίου Ρή προσωπική αυτή τη στιγμή. Εμεί μέχρι τι 7 Μαου θα πρέπει να καθορίσουμε την θέση μα, τη Επιτροπή μα δηλαδή. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ανάμεσα στι πολιτικέ ομάδε ούτε σε επίπεδο Επιτροπή. Ο Φρεντερίκ Νταρντέν έχει πρώτο το λόγο και ο κύριο Μπένιον στη συνέχεια. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχά την εισηγήτρια η οποία έρθε εδώ στην Επιτροπή μα για να μα δώσει τι πληροφορίε αυτέ όσον αφορά τα όσα συζητώνται στην Επιτροπή Προπολογισμών, στην οποία συμμετέχω και εγώ ως ένα πληρωματικό μέλος. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να κάνουμε και εδώ μια ανταλλαγή απόψεων. Θα αναφερθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, ποια είναι η δική μας η στάση. Σαφώς η κατάσταση είναι ιδιαίτερα λεπτή, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες, ιδίω όσον αφορά τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν για το 2013, ιδίω όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Επίσης, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα εγκριθεί ή όχι, με ποια μορφή και με ποια ποσά, με τι βαθμό ευελιξίας. Πολλοί λοιπόν οι αστάθμητοι παράγοντες και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις και συνδέονται τελικά και με τον ετήσιο προπολογισμό 2014 που συζητάμε εδώ. Άκουσα την παρέμβασή σας και όχι ως προς τη διαδικασία, αλλά ως προς την ουσία των πραγμάτων, βλέπω ότι είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα έλεγα και κάπως απεσιόδοξοι, καθότι λέτε ότι θα πρέπει ακόμα να εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις προπολογισμού ανταποκρίνονται στους στόχους μας. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την ε, βιωσιμότητα κάποιων ταμείων. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα μία αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν ακόμα και αν η χρηματοδότηση δεν τα αποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Δεύτερον, το χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι το ιδανικό χρονοδιάγραμμα το οποίο μπορούμε να εγκρίνουμε τη στιγμή που έχουμε τόσους πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Στα πλαίσια της έκθεσης του κυρίου Ορή εμείς θα κάνουμε κάποιες προτάσεις, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμα αυτά στη συνέχεια, όσο θα μας φτάνουν περισσότερες συγκεκριμένες πληροφορίες για όλα αυτά τα κρεμή ζητήματα. Δεύτερον, να σας θέσω και ένα ερώτημα. Αν δεν υπάρχει δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να έχουμε σημείο αναφορά στις οριακές τιμές 2013, ως προς τα ζητήματα τα οποία μας αφαιρούν εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Θα έχουμε τιμές οι οποίες θα είναι υψηλότερες, χαμηλότερες, μπορούμε να κάνουμε μια κάποια σύγκριση Ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα χωρίς ή με δημοσιονομικό πλαίσιο. Και διερωτάμε ιδιαίτερα όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πώς θα καταφέρουμε να εντάξουμε πολιετή προγράμματα απουσία πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και τι θα κάνουμε επίσης με το πρώτο έτος, με το πρώτο έτος χρηματοδότησης πώς θα καταφέρουμε να προωθήσουμε εμείς κάποια προγράμματα τα οποία καλύπτουν πολλά έτη. Τι θα κάνουν οι τοπικές οργανώσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα καταφέρουν να υποβάλουν προγράμματα και να ζητήσουν για αυτά χρηματοδότηση. Σε σχέση με κάτι που είπε ο κύριος Όρη, ζητήματα τα οποία εντάσσονται στη δική του τη έκθεση, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες για να προωθήσουμε κάποιες ε, πρωτοβουλίες όπως αυτή για την απασχόληση των νέων. Ήδη από την αρχή της περίοδου προγραμματισμού θα πρέπει να έχουμε χρηματοδότηση για την εγγύηση των νέων και θα πρέπει να καταφέρουμε να προωθήσουμε ταμείο όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, του οποίου καονισμός όπως είπατε αυτή τη στιγμή αναθεωρείται. Και βέβαια υπάρχει και το Ταμείο Προάσπισης των Απόρων που όπως είπε και η Πρόεδρός μας αυτή τη στιγμή συζητείται ακόμα η διάρθρωσή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε όμως και για το Ταμείο αυτό μια επαρκή χρηματοδότηση. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Yes, thank you. Um, firstly, um, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εγώ θα βασιστώ σε προτεραιότητες, γιατί όπως είπε και ο κύριος Ντάρμπιν, ο κύριος Ντάρμπιν μάλλον Μίλησε ήδη για τους ακαθόριστους παράγοντες του σταθεροποιητικού ταμείου. Τι λέει. Νομίζω λοιπόν θα περιοριστώ στις προτεραιότητες. Συμφωνώ γενικά με αυτά που είπε ο κύριος Ορή ως προτεραιότητες, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη και τους τομείς όπου μπορούμε όντως να κάνουμε κάτι και να κινήσουμε την οικονομία. Και κατ' εμέ το κυριότερο πρέπει να είναι η απασχολησιμότης των εργαζομένων. Η πρωτοβουλία απασχόληση των νέων ας πούμε πρέπει να στοχεύει αυτό ακριβώς την απασχολησιμότητα. Ίσως να μην μπορεί να δώσει βέβαια αμέσως δουλειές αλλά την απασχολησιμότητα τουλάχιστον να διασφαλίζει. Είναι ζωτικό να αρχίσει αυτό από τώρα και να μην περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Επίσης νομίζω πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης. είχα βάλει τροπολογίες για αυτό το θέμα και για την απασχόληση στην Ήπεθρο και για την εκπαίδευση των αγροτών καθώς και για το συνδυασμό των ειδικοτήτων για τους αγρότες. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και με τα χρήματα για τις κοινωνικές επενδύσεις και για τα περιφερειακά. Πρέπει δηλαδή να τονίζουμε πάντοτε ποιος θα είναι ο τύπος της εκπαίδευσης που χρειάζεται για να είναι απασχολήσιμος ο κόσμος και να έχει και κάποιο περισσότερο επιχειρηματικό πνεύμα. Δεν είναι το θέμα δηλαδή μόνο να μπορούν να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για τον ίδιο αριθμό θέσεων, αλλά να έχουν και τις ικανότητες να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν τεχνικά προβλήματα ως προς την υποστήριξη προγραμμάτων όπως εκείνο του Birmingham όπου υποστηρίζουμε την κοινωνική στέγαση μαζί με τη λήψη μέτρων ενεργειακής αποτελεσματικότητας γιατί έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας αλλά και περισσότερη αγοραστική δύναμη που κινεί την οικονομία. Γιατί υπήρξαν προβλήματα με τις επικαλύψεις και τους συνδυασμού προγραμμάτων και μπερδεύτηκαν τα πράγματα και με τις κρατικές ή μη επιχορηγήσεις. Αυτό να το προσέξουμε για να μην υπάρξουν επικαλύψεις και σταματήσουμε προγράμματα που πρέπει να συνεχίσουν και το αντίθετο ακόμη και για την επόμενη προγραμματική περίοδο να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι τα σωστά αυτά προγράμματα, τα πολύτιμα προγράμματα είτε πρόκειται για ομόλογα κοινωνικής απασχόλησης είτε όπως για να τα πούμε ότι θα μπορούν τα κράτη-μέλη να κάνουν την προσπάθεια να κινήσουν την οικονομία τους σε αυτές τις δύσκολες περιφέρειες. Και τέλος, έχω συναντήσει επιχειρήσεις και έχω θέσει ερωτήματα και α, έλαβα απαντήσεις. Τα τελευταία δέκα χρόνια λένε οι περισσότεροι γίνεται όλο και πιο δύσκολο και πιο γραφειοκρατική η πρόσβαση σε αυτά τα ταμεία και τα κονδύλια. Αν συνεχίσουμε να τα κάνουμε τα πράγματα δύσκολα Ίσως αυτό εξηγεί γιατί υπάρχουν ελλείψεις και δεν απορροφώνται όλα, δεν εφαρμόζονται πολλά προγράμματα. Γιατί δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να τα χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Καλώς. Κύριε Εισηγήτρια, ακούσατε ε, όλες αυτές τις αγορεύσεις ε, πώς μπορεί κανείς να έχει γνώμη για μια έκθεση που δεν υπάρχει σε ένα πολύ πλαίσιο που ακόμα δεν υπάρχει. κυρία Όρη, ε, τόση ώρα δεν μιλάγατε. Αμα μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, δύο στοιχεία ακόμα που λείπουν ακόμα από την παρουσίασή μου. Σύντομα, σύντομα. Τρεπετή, λέει ο κύριος Όρη στα γαλλικά. Ε, ναι, έχετε δίκιο λοιπόν κύρια Πρόεδρε. Το είπα και εγώ ο ίδιος. Προς το παρόν, απόψεις ανταλλάσσουμε για το πώς θα καταλήξουμε σε ένα συμβασμό ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, για τη βοήθεια προς τους απόρους ή τους πιο ε, αποκλεισμένους. Ε, τώρα συζητάμε για ένα ελάχιστο ποσό. Αυτή τη στιγμή είναι 3,5 δισεκατομμύρια και θα μειωθεί αυτό το κονδύλι. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε πολλά περιθώρια, ότι θα μειωθούν, γι' αυτό μιλούμε για ένα ελάχιστο ποσό. Και πάλι όλα αυτά είναι στα τυφλά. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε τα ποσά, ούτε πώς θα κατανεμηθούν, πώς θα γίνει ο προγραμματισμός μπορεί κάλλιστα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο κάθε χρόνο να ε, θέλουμε να υπάρχει κάποια διαφορετική στάθμιση. Δεν είναι στάνταρτα τα ποσά αυτά το ίδιο κάθε χρόνο. Αυτό είναι πρόβλημα. Πώς θα σταθμιστούν αυτά. Η πρόεδρος. Λοιπόν, ξέρετε ότι στην Επιτροπή μας εδώ το Λαϊκό Κόμμα επηρεάζει και τη σειρά ε, των αγορεύσεων μιλάει και στην αρχή και στο τέλος για να καταλαβαίνουμε καλύτερα. Έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε, κυρία Γιάντσεν. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση. Και όντως η δική σας Επιτροπή ασχολείται με συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα και το σημαντικό είναι πραγματικά να προχωρήσουν περισσότερο τα πράγματα, να προωθήσετε τα σημεία εκείνα τα οποία εσείς θέλετε να προωθήσετε στον δικό σας τον τομέα. Γιατί και οι ίδιοι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων έχουν πει ότι πραγματικά πρέπει να κάνουμε κάτι για την απασχόληση των νέων. Από ό,τι φαίνεται προ αυτό, στέλνουν ένα θετικό μήνυμα. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα το οποίο προωθούν και στα πλαίσια του προπολογισμού 2014, κατά πολέμηση της ανεργίας των νέων. Ως προς αυτό λοιπόν πρέπει να καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι τώρα εντοπίζετε το πρόβλημα και τώρα θα πρέπει να προωθήσουμε στεναρές λύσεις. Νομίζω ότι είναι εύκολο να το λέει αυτό κανεί, δύσκολο στη διαπραγμάτευση βέβαια. Τι θα γίνει αν δεν έχουμε πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Κοιτάξτε, ελπίζω ότι αν μη τι άλλο θα καταφέρουμε να έχουμε μια νομική βάση για τα διάφορα τμήματα του προπολογισμού. Γιατί στην περίπτωση αυτή θα έχουμε διαφορετικό πλαφόν, διαφορετική οριακή τιμή, η οποία όμω δεν διαφέρει τόσο πολύ για το 2014. Επομένως, δεν θα καθορίσει αυτό εντελώ τα πράγματα, αλλά και ω προ αυτό θα ήταν καλό να βρεθεί μια λύση. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ανταλλάσσουμε απόψει τότε και να κάνουμε διαπραγματεύσει. Α ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε αυτό. Μπορεί να ακούγομαι μερικές φορές λίγο απεσιόδοξη, αλλά πραγματικά ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση. Δεν θα είναι βέβαια αυτή η λύση που επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει αν μη τι άλλο να καταλήξουμε όσο το δυνατό περισσότερο σε μια καλή λύση. Ακόμα και αν το επίπεδο χρηματοδότησης τελικά είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο εμεί θέλουμε ή από αυτό που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας ελπίσουμε ότι τα ποσά τα οποία θα εγκριθούν τελικά θα μπορούν στην πράξη να απορροφηθούν. Όλοι οι προλύσαντες αναφέρθηκαν με μεγάλη σαφήνεια στις προτεραιότητές τους και αναφερθήκατε επίσης και στα διάφορα ζητήματα τα οποία προωθεί η Επιτροπή σας. Δεν αναφέρθηκα στις επιμέρους υπηρεσίες, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ξέρω ότι η δική σας Επιτροπή ασχολείται με τέσσερις οργανισμούς. Και αυτό το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά είναι ότι το Συμβούλιο κάνει περικοπές σε όλους αυτούς τους οργανισμούς, οριζόντιες περικοπές. Εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για τους οργανισμούς αυτούς ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα καταπολέμησης ανεργίας των νέων και όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Θα γίνει πάντως μια πρόταση προπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως σας είπα, και βάσει της πρότασης αυτής θα εργαστούμε και εμείς στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε λοιπόν με ιδιαίτερη μομονησία την δική σας πρόταση και στηριζόμαστε και σε εσά από την Επιτροπή Προπολογισμών προκειμένου να προωθήσετε και τα σημεία τα οποία εμείς προωθούμε εδώ στα πλαίσια της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για τον προπολογισμό 2014. Και ξέρω ότι ακούγεται κάπως ε, σουραλιστικό αυτή τη στιγμή ότι μιλάμε για το 2014, τη στιγμή που δεν έχουμε καθορίσει καν το πώς θα προχωρήσουμε με το ζήτημα του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και τις δημοσιονομικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω ότι θα έχουμε πάντως μια θετική πρόταση. Προχωράμε τώρα. Ερχόμαστε στην ε, πρόταση γνωμοδότηση του κυρίου Αρή ε, για την εντολή για το τριμερή διάλογο ε, για τον προπολογισμό του 2014 και ε, πραγματικά είναι πολύ ε, επίκαιρο. Κύριε Ισηγητά, έχετε το λόγο. Είμαστε στο σημείο 18, αν έχετε αντιληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ποιο τη χάρη μου σήμερα, λόγω μιλάω. Ε, ε, είμαι τυχερός. Πρέπει να σας πω ότι δεν πρόκειται να πω τίποτα άλλο. Διότι όλα αυτά που είπα προηγουμένως ε, παρουσία της κυρίας Γένσεν ε, συνοψίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και το σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης. Αν επιθυμεί τώρα η κυρία Πρόεδρος, μπορώ να επεκταθώ, ε, μπορώ και να επαναλάβω το όσο είπα, δεν έχω πρόβλημα. Πάντως, να θυμίσω ότι είναι σχέδιο γνωμοδότησης αυτό και η σημερινή είναι η πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων. Δεν ξέρω, ίσως προηγουμένως να μην τόνισα αρκετά την πρωτοβουλία για την νεολαία, για την απασχόληση των νέων, ούτε ανέφερα επαρκώς το θέμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Βοήθεια στους Απόρους. Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό. Έχουμε ακούσει ένα ποσό. Αυτό το ποσό πόθεν θα έρθει. Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από άλλη πηγή. Για να είμαι ειλικρινής, προς το παρόν ακόμα δεν είναι βέβαιο αυτό. Η πρόεδρος ήταν παρούσα. Στο Όσλο, όταν θέσαμε αυτό το ζήτημα υπόψη του αρμοδίου επιτρόπου. Ο οποίος σήκωσε τα χέρια του ψηλά και δήλωσε και αυτός άγνοια. Λοιπόν, σε σχέση με αυτή την εντολή για τον τριμερή διάλογο, ε, θα ήθελα να με υποστηρίξουν οι συνάδελφοι και ελπίζω οι δύο διαπραγματεύσει αυτές να ε, στεφθούν με επιτυχία και να ακολουθήσουν αυτή την ατραπό. Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο κύριος Ωρί, Νομίζω ότι αναφέρθηκαν κύριες προτεραιότητες και δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να προσθέσω για αυτό το θέμα. Θα καταθέσουμε λοιπόν μερικές τροπολογίες με επικοδομητικό πνεύμα για να βελτιωθεί αυτή η έκθεση. Α, πολύ ωραία. Ο κύριος Μπενιό. Και εγώ τόσο σύντομο θα προσπαθήσω να είμαι. Υποστηρίζω ιδιαίτερα την παράγραφο 3 για την απασχολησιμότητα των νέων ιδίω και την παραγραφό 4 για τη στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και την 7 για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως προ την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Και εμείς μπορεί να προσθέσουμε μερικές τροπολογίες, ιδιαίτερα για το θέμα της κοινωνικής στέγασης που λέγαμε, Γενικά όμως θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση και δεν βλέπουμε τίποτα που να, με το οποίο να διαφωνούμε ιδιαίτερως. Μάλιστα, δεν φαντάζομαι να θέλει να ξαναμιλήσει ο κύριος Ορή, όχι. Ε, τότε η διορία κατάσταση των προϊόν λίγη στις 17 Μαΐου το μεσημέρι. και θα τις εξετάσουμε στις 19 Μαΐου. και θα εγκριθούν στις 20 Ιουνίου. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα καταθέσει επισήμως την έκθεσή της, το σχέδιο έκθεσής της η κυρία Γιάνσεν. Ε, αυτά είναι περίεργα πράγματα. Εμείς οραθορίζουμε τη διορία των τροπολογιών για γνωμοδοτήσεις σε μια έκθεση που δεν ξέρουμε πότε. Επισήμως δεν την ξέρουμε. Τέλο πάντων, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, με τον όρο βέβαια μέχρι τότε να έχει κατατεθεί η έκθεση, γιατί αν στι 17 Μαου δεν υπάρχει το σχέδιο γνωμοδότηση τη κυρίας Γένσεν, τότε μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα είμαστε πιο ελεύθεροι. Λοιπόν, τέλο πάντων, παραμείνουμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα μέχρι να δούμε αν αλλάξει τίποτα αργότερα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στα πλαίσια της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Φτάνουμε στο 10 για το Ευρω... Ταμείο Ενίσχυσης των Απόρων. Για θέμα για το οποίο είμαστε στο εξή αρμόδιο. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να μας παρουσιάσει τις πιθανές συμβιβαστικές τροπολογίες Πρόκειται για έκθεση ναι. επί της οποίας δεχτήκαμε πολλές γραμματατήσεις Επιτροπή Προϋπολογισμών, Περίφ, Γεώρ, Πολίτ και Γίν και η συγγήτρια είχε πάει πάρα πολλές τροπολογίες 77 και συνέταξε 34 συμβιβαστικέ, 517 ήταν. Στο πολύ πρόεδρε, ιδιαίτερα τους σκιώδεις με τους οποίους συνεργάστηκα καθώς και το προσωπικό το δικό μου και όλων των πολιτικών ομάδων όπως είπε και η Πρόεδρος υπήρχαν 517 τροπολογίες και χρειάστηκε να τις εξετάσουμε πολύ γρήγορα αλλά καταλήξαμε σε 34 συμβιβαστικές. Τα κύρια θέματα που συζητήσαμε από τη συνεννόηση μας μέχρι τώρα ήταν τα εξής. Για την ομάδα στόχευσης Ορισμένες τροπολογίες πρότειναν την παράταση, την επιμήκυνση, τη διεύρυνση αυτής της ομάδας, αλλά επειδή δεν υπήρχαν τα απαραίτητα κονδύλια, τα 2,5 δισεκατομμύρια σε 7 χρόνια δηλαδή και επειδή αυξάνεται η ανέχεια σε ολόκληρη την Ένωση από τότε που άρχισε η κρίση και βλέπουμε πόσοι χρειάζονται να καταφύγουν σε τράπεζες τροφίμων και κοινωνικά παντοπολία καθώς και στην ε, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα βλέπουμε ότι οι τράπεζες τροφίμων έχουν γίνει πολύ χρήσιμες. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα τους πιο φτωχούς και εκείνους που χρήζουν περισσότερης βοήθειας, εκείνους που δεν έχουν τα απαραίτητα τρόφιμα δηλαδή και πρόκειται για το μόνο πρόγραμμα που στοχεύει αυτούς τους ανθρώπους. Ως προς το εύρος τώρα, γενικά υποστηρίχθηκε η ιδέα να υπάρξει με ευρύτερο εύρος, ευρύτερο εύρος λέγω, και πεδίο εφαρμογής. Ακούσαμε και μη κυβερνητικέ οργανώσεις που μας είπαν ότι προτιμούν να διευρυνθεί το πεδίο τουλάχιστον για τη βασική ηλική βοήθεια πέρα από τη βασική ηλική βοήθεια γιατί αυτήν τη χορηγούν ήδη οι ΜΚΟ Οι συμβιβαστικές τροπολογίες ε, αφήνουν το θέμα αυτό του εύρους στις χώρες μέλη για την διατροφική ή και υλική βοήθεια. Ως προς τη χρηματοδότηση των προϋπολογισμών του προγράμματος, γενικά υπάρχει συμφωνία ότι τα 2,5 δισεκατομμύρια δεν επαρκούν. Αυτό μας ανησυχεί διότι τα πράγματα είναι όλο και πιο δύσκολα και δεν θα αρκέσει για τίποτα. Οι διαπραγματεύσεις για το MFF, στις διαπραγματεύσεις για το MFF και η πρόεδρός μας και ο κύριος Λαμασούρ έστειλαν επιστολές ζητώντας αύξηση σε 3,5 δισεκατομμύρια με πλήρη δικαιολόγηση και επιστολή και από την, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Υπήρξαν πολλές τροπολογίες για το θέμα της χρηματοδότησης και συζητήσεις που κατέληξαν στο ότι καλύτερο ήταν να παραμείνει η αρχή πρόταση της Κομισιόν 85% χρηματοδότηση με τις κανονικές συνθήκες και ιδιαίτερη κατά 90-95% για τις χώρες στόχευσης. Έγιναν επίσης πολλές συζητήσεις για να δούμε αν το πρόγραμμα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή εθελοντικό. Η δική μου θέση ήταν ε, εκείνη της Κομισιόν να είναι υποχρεωτικό για όλες τις χώρες μέλη δεσμευτικό ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο βοήθεια αλλά κατατέθηκαν τροπολογίες από όλες τις πολιτικές ομάδες που ζητούσαν εθελοντική συμμετοχή. Το θέμα συζητήθηκε τέσσερις φορές σε συναντήσεις των σκιωδών και ακούστηκαν πολλές, πολλά αιτήματα για εθελοντική συμμετοχή από πολλές ομάδες. Ακόμη όμως συζητιέται αν πρέπει να γίνει υποχρεωτικό ή όχι. Επομένως καταλήξαμε ότι εάν το πρόγραμμα είναι εθελοντικό τότε πρέπει να κρατηθεί παρόλα αυτά κάποιο ποσό στον προϋπολογισμό μέχρι να αποφασιστεί αυτό. ή για να υπάρχει δυνατότητα να συνδυαστεί και με άλλα ενωσιακά προγράμματα όπως της διατροφικής βοήθειας. Πολλές επίσης ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις δέχονταν την ιδέα και συνοδευτικών μέτρων μια γαλλική οργάνωση είπε ότι 75% των ε, ανθρώπων που αποφελούνται από την οργάνωση δεν θα επιστρέψουν για δεύτερη χρονιά γιατί ο στόχος είναι να μπορέσουν να περάσουν από το πρόγραμμα αυτό σε άλλα ενωσιακά προγράμματα. Έχουν επίσης ακουστεί αρισμένες ανησυχίες ως προς τη μετάβαση, τη μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, αν είναι θελοντική συμμετοχή, τότε με τη συμφωνία και του MFF πρέπει να γίνει μία ομαλή μετάβαση από τα υπάρχοντα προγράμματα στο καινούριο το 2014 και ζητήθηκαν λοιπόν μεταβατικά μέτρα. Γι' αυτό συγγράψαμε μία συμβιβαστική που τονίζει την ανάγκη για αυτήν την ομαλή μετάβαση. Άλλα βασικά θέματα των συμβιβαστικών τροπολογιών είναι η ενδυνάμωση της ε, εταιρικής ε, σχέσης όσων θα συμμετάσχουν και η διαφάνεια. Επίσης μιλήσαμε για τα υγιή τρόφιμα και για την αποφυγή του στιγματισμού όσων θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα. Τονίσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει άχρηστη πρόσθετη γραφειοκρατία ή διοικητικών άχθος γιατί στόχος μας είναι να διευκολυνθεί η λειτουργία των μήκη όμικρων. Τέλος υπήρξε μεγάλη συνένεση ότι δεν πρέπει να είναι αυτό το μόνο ενωσιακό εργαλείο για την καταπολέμηση της ανέχειας, αλλά απλώς ένας μοχλός διευκόλυνσης. Δεν κερδίζετε καθόλου χρόνο μιλώντας τόσο γρήγορα, λέει η Πρόεδρος, γιατί δεν μπορούν να σας παρακολουθήσουν οι διερμηνευτέ. Ούτε τα μισά δεν μεταφράζονται. Α, με συγχωρείτε, συγγνώμη και στους διερμηνευτάς. Ας καταλήξω λοιπόν. Αν έχουν τα μέλη καμιά απορία mm. ως προς τα γενικό, τις γενικότερες αρχές που ανέφερα, ή μάλλον για να επαναλάβω, το πρόγραμμα αυτό το feed είναι συμπληρωματικό των υπολείπων εργαλείων και μέτρων για την καταπολέμηση της ανέχειας. Αλλά είναι από τα σημαντικότερα για το θέμα αυτό που σας είπα της καταπολέμησης της ανέχειας στην Ένωση. Ώστε να διευκολυνθεί η ζωή 20 εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Ευχαριστώ τους Κιώδης, συναντηθήκαμε πέντε φορές και υπάρχει κι άλλη συνάντησή μας που βλέπετε αυτή την εβδομάδα για να τελειώσει η εξέταση των συμβιβαστικών που πρωτοϋποβλήθηκαν σήμερα και επειδή δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο ζητήσαμε να αναβληθεί η ψηφοφορία για τις 7 Μαΐου αντί για αύριο. Τέλος, η Ιρλανδική Προεδρία θεωρεί το πρόγραμμα προτεραιότητά της και ο πρόεδρος του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ Τζον Μπάρντεν συνεργάζεται μαζί μας και ελπίζω να συνεργαστώ με την Ιρλανδική Προεδρία και με τους σκιώδεις και γενικότερα ώστε να καταλήξουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τελεία. Μάλιστα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα σας πω ποιοι είναι για να μου πείτε αν συμφωνείτε. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να δώσω δύο-τρει φορέ το λόγο στου ίδιου συγητέ αυτή τη στιγμή, στους ίδιου ομιλητέ. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δώσω επίτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μπορούμε να μιλήσουμε πάρα πολύ ώρα γιατί θα έρθει η Επίτροπος Βασιλείου στι 5.30. Δυόμιση λεπτά ο καθένας. Ξεκινάμε με τον κύριο Τομασμάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι καταρχάς που εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης φέρουμε αυτή την ευθύνη ε, καθήλυνα αρμόδια και όχι η Επιτροπή Γεωργίας. Ήταν ένα πρόγραμμα επισητισμού ε, δωρεάν παροχή τροφίμων και αυτό ήταν λέει στην Επιτροπή Γεωργίας. Όχι, καλό είναι στη δική μας Επιτροπή. Γιατί εμείς θέλουμε να δούμε πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα. Να πούμε ότι ένα ε, λογικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης της στόχης είναι κάτι στο οποίο να συνεργαστούμε κι εμείς. Και χαίρομαι για τη συνένεση που πριτάνευσε μεταξύ των σκιωδών για την αύξηση των πόρων. Η Κομισιόν πρότεινε 2,5 δις, εμείς προτείναμε 3,5 δις. Αύξηση κατά 1 δισεκατομμύριο. Είναι σημαντικό αυτό αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε ένα πρόγραμμα ε, το οποίο είχε τεθεί στην αρχή. 100% όχι. Είπαμε, συγχρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρηθεί και σε όλα τα άλλα προγράμματα που έχουμε, όλα αυτά είναι συνυπευθυνότητα. Ε, φέρουν ευθύνη και τα κράτη-μέλη. Βρέθηκε λοιπόν μια τέτοια ρύθμιση, 85% ε, στην κανονική κατάσταση και 95% σε χώρες που ακολουθούν προγράμματα και μνημόνια. Ε, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα πραγματικά πραγμα καταπολέμησης της φτώχειας να καταλάβουν ότι δεν είναι πρόγραμμα αυτό υποκατάστασης, αλλά συμπλήρωσης. Ε, σε πολλά κράτη-μέλη λειτουργεί αυτό, αλλά σε ορισμένα δεν το προωθούν καθόλου. Θα ήθελα να πω, κυρία Κοστέλο, και να τονίσω και πάλι, ότι είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και υποχρεωτική η αναφορά ε, και η καταγραφή. Αυτό το έχουμε εξασφαλίσει. Για μένα είναι σημαντικό. Βεβαίως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τα καθήκοντά τους. Δίνουμε κι εμείς ε, το μερίδιο που μας αναλογεί, τσοντάρουμε δηλαδή, αλλά ε, θα πρέπει τα κράτη-μέλη με ένα απλό τρόπο να τα εφαρμόζουν για να μπορούν να εφαρμόζουν. Αλλιώς υπάρχουν αντιστάσεις στα κράτη-μέλη που λέγουν ότι γίνεται τεράστιος χαμός για τόσο λίγα χρήματα. Θα πρέπει να είναι απλά ε, τα πράγματα για να μπορούμε να έχουμε λογική εφαρμογή και αποτέλεσμα σε τελική ανάλυση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα έχετε καταφέρει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ο Φιλ Και μετά η κυρία Σρόη. Ah, uh, um, Σας ευχαριστώ. Μιλώ αυτή τη στιγμή εξ ονόματος της Μάριον Χόκκιν, η οποία δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την εξαιρετική συνεργασία που είχαν για την έκθεση αυτή. Και ουσιαστικά λέει ότι υπάρχουν κάποια σημεία συμφωνίας για όλες τις συμβαστικές τροπολογίες, εκτός από την τροπολογία για το άρθρο 6 Έπειτα, οι ε, φιλελεύθεροι δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να συμπεριληφθούν κάποια αριθμητικά δεδομένα τα οποία θα αποτελούσαν αύξηση για τη γραμμή του προπολογισμού. Αυτό συνάδει και με ε, άλλα νομοθετικά κείμενα τα οποία έχουν να κάνουν με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υποστηρίζουμε να έχει εθελούσια ο χαρακτήρα το ταμείο αυτό, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί ουσιαστικά να ξεμπλοκάρει αυτή η μειονότητα που μπλοκάρει τώρα την πρωτοβουλία αυτή. Επίσης, όσον αφορά το άρθρο 2, υποστηρίζονται οι προτάσεις για την απλούστευση του Ταμείου, σε σχέση με τον εθελούσο χαρακτήρα του Ταμείου τώρα. Και τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν τα χρήματα από τα κράτη-μέλη, που συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν τελικά στο Ταμείο, η Επίτροπος μας είχε πει στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα ότι μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα όπου τα χρήματα τελικά θα είναι διαθέσιμα για το Ταμείο αυτό. Συμφωνούμε επίσης με τη συγχρηματοδότηση αρκεί να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και το Ταμείο Συνοχής. Επειδή έχει μετατεθεί ψηφοφορία, έχουμε πλέον περισσότερο χρόνο για να επιλύσουμε κρεμή ζητήματα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ελιζαμπέθ θα μπορώ να είμαι πολύ συντομή, διότι η Σκιώδης, ε, η συγκήτρια κυρία Κονέλησεν ενήρθε. Κατά την άποψή μου, υπάρχουν κάποια σημεία ε, που με αφορούν, γιατί ε, εργάζομαι στην πρόταση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο συμβατό με το Κοινωνικό Ταμείο, το ιδεώδες να το χειρίζει το ίδιος οργανισμός σε κάθε χώρα, γιατί έτσι θα βγει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Από ό,τι φαίνεται αυτό δεν επετεύχθη. Εν πάση περιπτώσει να είναι ήδη οι κανονισμοί και, του, και οι μηχανισμοί μάλλον ε, και να υπάρχει δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να το αναθέσουν στην ίδια διοικητική υπηρεσία. Ε, επίσης, το θέμα του εθελοντικού χαρακτήρα είναι για μας το σημαντικότερο, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν άλλες λύσεις και δεν χρειάζονται ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γιατί έχουν τα δικά τους, τοπικά, εγχώρια προγράμματα. Και επειδή τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι. Αφήστε που είναι πολύ λίγα τα λεφτά και πολλά τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υποφελούνται εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να μην προσθεθούν και άλλα κράτη, γιατί θα μειωθεί το ποσό. Ε, που τους αναλογεί. Ε, χαίρομαι λοιπόν για αυτό τον εθελοντικό χαρακτήρα. Επίσης χαίρομαι και θεωρώ σημαντική τη χρηματοδότηση. Συγχρηματοδότηση είναι αυτή, γιατί ε, αυτή απαιτείται για να υπάρχει και δημοσιονομικός κανονισμός, αλλιώς δεν θα ήταν επιτρεπτή αυτή η στήριξη στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου την εισηγήτρια για την εργασία που έχει κάνει και για τον νέο ορισμό του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας. Νομίζω ότι το πεδίο εφαρμογή αυτό είναι καλό. Τώρα να μιλήσω και εγώ για τον θελοντικό χαρακτήρα του Ταμείου. Το είπε η εισηγήτρια ότι δεν έχουν συμφωνήσει αυτή τη στιγμή οι πολιτικέ ομάδε και έχουν υποβληθεί πολλέ αντιφατικέ τροπολογίε για το ζήτημα αυτό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακολουθούν οι συνάδελφοι αυτόν τον δρόμο. Ήδη κάναμε τη συζήτηση αυτή όταν εγκρίναμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και ορισμένα κράτη-μέλη κατά την έγκριση στρατηγικής αυτής είχαν πει ότι η μαϊένδια, η φτώχεια δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ζήτημα επικουρικότητας, είναι καθαρά εθνικό ζήτημα. Και αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα είναι ότι αυξάνεται η ένδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακούω το ίδιο επιχείρημα αυτή τη στιγμή από ορισμένα κράτη-μέλη που θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά εγκρίνοντας την εγγύηση για την νεολαία έχουν καλύψει όλο το κοινωνικό τους κομμάτι, όλες τις κοινωνικές υποχρεώσεις τους και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα παραπάνω. Μα δεν είναι αυτό η Ευρωπαϊκή Ελληνική όμως. Επειδή ορισμένοι κινητοποιούν τις εκκλησίες τους για να βοηθήσουν τους άπορους, δεν μπορούν να λένε αυτή τη στιγμή ότι δεν θέλουν να υποστηρίξουν παράλληλα και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθηθεί μια ευρωπαϊκή ελληνική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρωπαϊκό μήνυμα. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, σφάλουμε πάρα πολύ. Επίσης, αν δεν προωθήσουμε το Ταμείο αυτό, ουσιαστικά αντιβαίνουμε στα όσα λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν εγκρίναμε ένα σχετικό ψήφισμα με 540 ψήφους υπέρ, με ελάχιστε ψήφους κατά και ελάχιστες αποχές. Και θυμάστε ότι στα συμπεράσματά μας είχαμε πει ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε τους πιο άπορους ανθρώπους και ότι θέλουμε να δώσουμε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και ουδέποτε λέγαμε στο ψηφισμά μας ότι θα έχει θελούσιο χαρακτήρα το ταμείο αυτό, αυτή η χρηματοδότηση. Και τέλο, βλέπω ότι ορισμένα κράτη-μέλη μένουν στη θέση του. Ενδεχομένω να πρέπει να είναι εθελοντικό ο χαρακτήρα του Ταμείου αυτού. Προτού όμω καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτό, θα πρέπει να μα δοθούν κάποια εχέγγυα για το πώ θα επηρεάσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για το πώ θα επηρεάσει το Γενικό Προπολογισμό. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε προωθώντα το Ταμείο αυτό και λέγοντα ότι εξ αρχή θα πρέπει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Ας σκεφτούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, ακόμα και η δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ακόμα και ορισμένα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι άδικο το γεγονός ότι συμμετέχουν μόνο ορισμένα κράτη-μέλη και όχι άλλα. Επομένως, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει επίσης και αν βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο αυτή τη στιγμή, προτού καταλήξουμε τελικά και εμείς τη δική μας ψηφοφορία. Πρώτα όμως να δώσω το λόγο στον κύριο Ορή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για την εργασία αυτή την οποία έκανε. Ιδιαίτερα ουσιαστική. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες εντάσεις. Είναι και ιδιαίτερα όμως διαλλακτική και γι' αυτό την ευχαριστώ. Την ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ καλή συνεργασία και για τον συντονισμό που εξασφάλισε στα πλαίσια της συνεργασίας μας. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στις 7 Μαΐου, γιατί δεν είχαμε ακόμα αρκετό χρόνο για να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία για όλα τα σημεία της έκθεσης. Αυτή τη στιγμή η παρέμβασή μου έχει ένα διτό χαρακτήρα. Καταρχάς, Ξέρετε ότι είχαν ε, εκφραστεί κάποιες επιφυλάξεις, ακόμα και φόβος θα έλεγα, όσον αφορά το επιστημιστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους απόρους και από την άλλη βλέπουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα ταμείο ενίσχυσης των απόρων. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά η διαδικασία απλουστεύεται κατά αυτόν τον τρόπο και όλη η διαθέσιμη χρηματοδότηση τελικά θα πάει στους πιο άπορους και όχι, και όχι στην διαχείριση του ταμείου. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει συγχρηματοδότηση, γιατί μιλάμε εδώ πέρα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επιβάλλεται λοιπόν η συγχρηματοδότηση. Προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη λύση προκειμένου να μεταπίσουμε κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να προωθήσουν την πρότασή μας. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές στο παρελθόν αναφέρθηκα στα εθνικά προγράμματα, στα εθνικά επιδόματα. Τώρα, είτε έχει θελοντικό είτε έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα το πρόγραμμα αυτό, το σημαντικό να καταλάβουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία τονίσατε και εσείς κυρία Πρόεδρε και τα οποία σχετίζονται και με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Πάντως, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η αρμοδιότητα είναι καθαρά εθνική. Και εφόσον μιλάμε για εθνική αρμοδιότητα, ακόμα και αν το ζήτημα αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ακόμα και αν εμείς ψάχνουμε εδώ πέρα λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρμοδιότητα παραμένει κυρίως εθνική. Νομίζω ότι θα πρέπει να δαπανούμε λιγότερα ποσά στην διοίκηση, στην διοικητική διαχείριση και θα πρέπει να δίνουμε τα χρήματα αυτά στους απόρους. Είχαμε δει στο παρελθόν ότι ακόμα και τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ δεν φτάνανε. Τι θα κάνουμε τώρα με τα 2,5 δισεκατομμύρια, το μικρό αυτό ποσό με το οποίο έχουμε καταλήξει. Πολύ φοβάμαι ότι περιπλέκουμε πάρα πολύ τα πράγματα και ξεχνάμε την ουσία ότι αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ελάχιστα τελικά και αν μη τι άλλο θα πρέπει να φτάσουν στους τελικούς δικαιούχους. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σεν και μετά ο κύριο Σέρκα. Yeah, Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πραγματικά κάνει εξωθαύμαστη δουλειά και είναι τεράστιε ε, οι τροπολογίε, ο αριθμό του δηλαδή. Προσπαθήσαμε και τη μειώσαμε. Ε, έχουμε ακόμα κάποιε διαπραγματεύσει παρόλο που έχουμε δαπανίσει ε, ώρε επί ωρών σε διαπραγματεύσει, επικοδομητικέ και ενδιαφέρουσε δεν λέω. Ε, το ένα θέμα είναι ακριβώς αυτός ο εθελοντικός σημεί χαρακτήρας. Η μεγάλη ε, πλειονότητα πιστεύει ότι θα πρέπει να παραμείνει εθελοντικό το πρόγραμμα, να δούμε ποιο τρόπο θα βρούμε για να το εφαρμόσουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Ρή ότι παρόλο που όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναγκαστούν να καταπολεμήσουν την φτώχεια. Δεν είναι, πρέπει σώνει και καλά να γίνει μέσω αυτού του προγράμματος, αυτού του ταμείου. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν θέλουν να δαπανίσουν κρατικά κονδύλια για άμεση επισητιστική βοήθεια και συσίτια, εν πάση περιπτώσει. Τα προγράμματα αυτά Ε, δεν θα πρέπει να σταματήσουν ξαφνικά γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εξαρτώνται για την ε, επιβίωσή τους ε, από τα τρόφιμα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα πρέπει όμως τα χρήματα αυτά να χαθούν και να πάνε στο γενικό προϋπολογισμό. Τώρα, κάτι που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ ως προσθήκη για το Ταμείο είναι να μπορεί να χρησιμοποιείται για πιο μικρή διατροφική αλυσίδα ε, από ντόπια τρόφιμα και να μην έχουμε σπατάλες ε, τροφίμων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο πετάμε 90 εκατομμύρια τόνους τροφίμων. Τα 20 από αυτά είναι πολύ υγιεινά και κατάλληλα προς κατανάλωση η Ουγγρική Επιστημιστική Τράπεζα, η Τράπεζα Τροφίμων, το τόνισε αυτό και νομίζω ότι έτσι δεν τους δίνουμε μόνο ψάρια, αλλά τους μαθαίνουμε να ψαρεύουν ε, για να μην πετάμε τρόφιμα πολύτιμα και υγιεινά και ταυτόχρονα να κερδίζουν και κάποια ανεξαρτησία, να απεξαρτηθούν από το πρόγραμμα ε, οι οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τελικά θα μπει και στην πρόταση. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σέρκας και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι ο λεγόμενος εντός εισαγωγικών εθελούσιος χαρακτήρας του προγράμματος. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί κάποιοι συνάδελφοι υπέγραψαν τροπολογίες ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση Πίσω από τον εθελοντικό ή χαρακτήρα εδώ τι κρύβεται. Άλλη συζήτηση. Όχι για το ε, αν θέλει κάποιος να συμμετέχει. Μα έτσι και η συμμετοχή στα προγράμματα είναι εθελοντική, δεν τον αναγκάζει τον άλλο να το χρησιμοποιήσει. Και το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και όλα τα υπόλοιπα. Δεν σου βάζει κανεί το μαχαίρι στο λαιμό. Εδώ άλλα συζητάμε, Πρόεδρε. Τα λεφτά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλου σκοπού. Αυτό συζητάμε. Υπάρχουν κράτη-μέλη που θέλουν να πάρουν αυτά τα λεφτά, λέει, για τους απόρους, για τις τράπεζες ε, τροφίμων και μετά τα, βάζουν σε αυτοκινητοδρόμους ή σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, πίσω από τον εθελοντικό χαρακτήρα θα αφήσουμε τα κράτη-μέλη να λονίζουν με χρήματα που είναι για τους απόρους να τα ε, χρησιμοποιούν ε, για αλότριους σκοπούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει αν θα μπει ο εθελοντικός χαρακτήρας στην γνωμοδότηση δεν με νοιάζει να μπει αυτό, απλώς να χρησιμεύει μόνο για τα θέματα των απόρων. Αυτό είναι το πεδίο εφαρμογή και όχι γενικά πάρτε τα. Αν δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να ανατρέξουν, με γεια τους με χαρά τους, αλλά όχι να τα πάρουν και να τα δώσουν αλλού. Γιατί τελικά, όπως συμβαίνει πάντα, χρησιμοποιούμε κάποιες λέξεις για να συγκαλύπτουμε ή να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα. Εθελοντικό θα είναι, αλλά όχι να πάρουν τα λεφτά από τους απόρους, να τα βάλουν σε αυτοκινητοδρόμους οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Και θα πάρουμε του φτωχού ταρνί και θα το κάνουμε αυτοχειρητόδρομο Ή οτιδήποτε, δεν ξέρω εγώ, εκπαίδευση, κατάρτιση, όχι. Αυτά τα λεφτά είναι για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν ούτε να φάνε, ούτε να στεγαστούν, ούτε να ντυθούν, ούτε να ζεσταθούν, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το ζήτημα και οι συνάδελφοι που έχουν κάνει προπολογίες για τον εθελοντικό χαρακτήρα, δεν λέω καλοπροαίρετα, ε, και ε, ε, δεν θα πρέπει να τους χειραγωγούν κάποιοι κακοπροαίρετοι και κάποιοι που θέλουν να σφετεριστούν αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα της ανασχετικής ε, στο Συμβούλιο που μπλοκάρει. Ναι, αλλά τι θα γίνει, δεν θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Δεν χρειάζεται Δηλαδή, αμαχητή, θα προχωρήσουμε, θα μα επιβάλλουν τον κανόνα. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά έχει φτάσει η Επίτροπο και περιμένει έξω από την πόρτα. Mm. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει τώρα για αυτό το θέμα. Θα είμαι πολύ σύντομη. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπαν οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση αυτή, η πρόθεσή της ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τις περισσότερες ανάγκες, τους πιο ευάλωτους δηλαδή, και οι οποίοι δεν είναι δικαιούχοι άλλων προγραμμάτων. Αυτό είναι το βασικό πνεύμα της πρότασης αυτής. Δεν νομίζουμε ότι έχει να κάνει με ανακατανομή ή με αναδιοργάνωση των διατηθέμενων ποσών. Νομίζω ότι έχουμε προτείνει ένα σύστημα εφαρμογής και ένα σύστημα προγραμματισμού το οποίο είναι απλό, εύκολο στην εφαρμογή του. Παρακολουθούμε λοιπόν εκ του σύναγκη σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται προκειμένου να καταφέρουμε να πλουστεύσουμε το σύστημα αυτό ακόμα περισσότερο. Σας διαβεβαιώ πάντως ότι ε, διατηρούμε τις ευθύνες μας όσον αφορά την ε, χρηστή διαχείριση της κοινοτική χρηματοδότησης. Αυτό αποτελεί μία από τις βασικές αρχές του συστήματος αυτού. Και τέτοια τα κράτη-μέλη οργανώνονται από μόνα τους για το πώς θα διαθέτουν τα ρούχα, τα τρόφιμα, προκειμένου πραγματικά να φτάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους δικαιούχους, να υποστηρίξουν στην ουσία αυτούς τους ανθρώπους. Για μας η πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειρίας είναι ένα πολύ καλό μέσο, ακριβώς επειδή υπάρχουν ευέλτιστες πρακτικές ορισμένα κράτη-μέλη, τις οποίες θα έπρεπε να γνωρίζουν και άλλα κράτη-μέλη και άλλοι φορείς, δημόσιοι, ιδιωτικοί, οι οποίοι εμπλέκονται ιδιαίτερα στην υποστήριξη των απόρων και θεωρούμε ότι το ταμείο αυτό ουσιαστικά αν εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη θα προωθήσει περισσότερο και τον σχετικό θελοντισμό στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε. Η συγγήτρια έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους καθώς επίσης και για τις περαιτέρω τροπολογίες που υποβάλλουν για την πρόταση αυτή και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποστήριξή της. Απαντώντας τώρα σε ορισμένες παρεμβάσεις. Όντως, με την ε, εξαίρεση ορισμένων σημείων μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που ο κύριος ε, Μπένιαν ότι όντως θα πρέπει να αυξηθεί χρηματοδότηση σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια ενός ευρύτερου πεδίου εφαρμογή και εφόσον συμμετέχουν περισσότερα κράτη-μέλη. Κύριε Μαν, Όντω και εμεί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απλουστευτεί περισσότερο το σύστημα και όπω είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύστημα ανταλλαγή εμπειριών ακριβώ αυτό προσβλέπει και παράλληλα προσβλέπει ότι υπάρχει ένας καλύτερος έλεγχος. Από τη συζήτηση που έγινε σήμερα το απόγευμα βλέπω ότι ένα ακαθόδε ζήτημα είναι ο θελοντικός ή μη χαρακτήρας του Ταμείου. Όπως είπε ο κύριος Σέρκας, η βασική ιδέα είναι τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή να καταλήξουν τελικά στους πιο ευάλωτους ανθρώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και αύξηση του ποσού αυτού εφόσον γίνεται αλλά πάλι οτιδήποτε ποσό και αν εγκρίνουμε θα πρέπει να πάει στους τελικούς δικαιούχους. Οι συμβαστικές τροπολογίες, οι σχετικές με το ποσό, έχουν να κάνουν με τα ζητήματα αυτά, ιδίως με το ζήτημα της συμμετοχής Ξέρω όμω ότι έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά τουλάχιστον μέχρι τι 7 Μαου θα πρέπει να καταφέρουμε να διευθετήσουμε τα εκκρεμή ζητήματα και να έχουμε τελικά μια ικανοποιητική συμφωνία, ένα ικανοποιητικό συμβασμό μέχρι τι 7 Μαου που θα γίνει και η ψηφοφορία. Σα ευχαριστώ και πάλι. Μέχρι τις 6 ε, Μαΐου στις 4 το απόγευμα θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι συμβαστικές τροπολογίες και θα ψηφίσουμε σε 7 Μαΐου. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό της μερίσιας διάταξης και κάνουμε μια σύντομη διακοπή για να υποδεχθούμε την Επίτροπο.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 Euh, Κυρία Επίτροπε, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε, θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Θελήσαμε να σας καλέσουμε τη στιγμή όπου συζητιέται η πρωτοβουλία σας «Έρασμος για όλους». Και που αποτελεί πρόγραμμα που ανταποκρίνεται σε, στις επιτυχίες της Ένωσης. Σήμερα συνεργάζεστε με τον Επίτροπο Λάσλο Άντορ για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Κομισιόν υπέρ των νέων. Στην ενδιάμεση αυτή περίοδο, στο ενδιάμεσο αυτό πλαίσιο μεταξύ παιδείας και ανάληψης εργασίας. Κάτι έπρεπε να κάνει λοιπόν η Ένωση και γι' αυτό. Ξέρετε ότι η Κομισιόν έχει αναλάβει δεσμεύσεις από αυτού. Και εμείς σήμερα συζητήσαμε τις τροπολογίες που θα εγκρίνουμε για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και εξετάζουμε έκθεση που καλύπτει ορισμένες πτυχές από τη δική σας πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερα και σας δίνω μέσω στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και για μένα είναι μεγάλη η η παρουσία μου εδώ μπροστά σας. Κυρίες και κύριοι, φέτος το Φεβρουάριο πάνω από 26 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρέθηκαν χωρίς δουλειά δηλαδή ρυθμός ανεργίας 12%. Η σοβαρότερη ανησυχία μας είναι η κατάσταση των νέων. Περίπου 5,7 εκατομμύρια είναι άνεργοι. Κοινωνικά αυτό είναι, δεν είναι βιώσιμο και ηθικά είναι απαράδεκτο. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είναι βέβαια μία από τις κύριες τους κύριους λόγους για την ανεργία στην Ευρώπη σήμερα. Όσο παραμένει χαμηλή η ανάπτυξη, οι θέσει εργασία θα είναι λιγοστέ. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλοι τι πόρους διαθέτουμε για να προσφέρουμε πραγματικές λύσεις στους νέους, αλλιώς θα υπάρξει ακόμη μια χαμένη γενιά. Γι' αυτό υπό την ηγεσία του συναδέλφου μου Λάσλο Άντορ, η Κομισιόν πρότεινε την νεανική εγγύηση. Χαίρομαι γιατί και μετά το ψήφισμά σας το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου κατέληξε σε μια συμφωνία για τη σύσταση για τις εγγυήσεις των νέων που ανοίγει το δρόμο για δράση από τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν ώστε να βοηθήσουν τους νέους. Αλλά για να λυθεί το ενδημικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων η παιδεία και εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση, η επαγγελματική μετεκπαίδευση είναι κεντρικά θέματα σε στιγμή μάλιστα που ο κόσμος ζητάει γρήγορες λύσεις για οξία προβλήματα. Ξέρουμε ότι η παιδεία είναι πάντοτε μακροπρόθεσμο θέμα και που φέρνει καρπούς στο τέλος μόνο της διαδικασίας. Παρ' όλα αυτά είμαστε πεπισμένοι ότι είναι το κλειδί και για την άμεση ανταπόκριση που πρέπει να δώσουμε στην κρίση. Βοηθώντας τον κόσμο να βρει δουλειά και βελτιώνοντας την αποσχολησιμότητά τους. Ας είμαστε σαφείς. Η δημόσια εκπαίδευση παραμένει από τα καλύτερα εργαλεία για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζω και εγώ ως αρμόδια επίτροπος για την παιδεία. Πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο για να οπλιστούν οι νέοι με το σωστό μείγμα γνώσης και δεξιοτήτων παρά την υψηλή ανεργία, ο αριθμός των κενών θέσεων αυξάνεται επίσης. Πάνω από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις υπάρχουν στην Ευρώπη και αυτό είναι απαράδεκτο παράδοξο. Διότι δείχνει πάνω απ' όλα ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων που χορηγούνται και των αναγκών του κόσμου της εργασίας και σε κάποιο βαθμό και την αποτυχία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μέχρι το 20 αναμένουμε ότι 36% όλων των θέσεων απασχόλησης στην Ένωση θα απαιτούν υψηλές δεξιότητες. Σήμερα μόνο 26% του εργατικού μας δυναμικού έχει φτάσει σε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη και αν ισχύει παρά το ότι ισχύει ότι και οι όσοι έχουν υψηλή μόρφωση επίσης πλήττονται από την κρίση, η εμπειρία δείχνει ότι αυτοί έχουν καλύτερη τύχη από τους άλλους. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι περισσότεροι νέοι θα φτάνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι και το νόημα του στόχου για την Ευρώπη 2020 που έχουμε θέσει. Η Ευρώπη χρειάζεται ανθρώπους με τη γνώση και τη δεξιότητα για να καθοδηγήσουν να επιτύχουν την ανάπτυξη. Σήμερα όμως οι εταιρείε δεν τους βρίσκουν, δεν δεν παράγουμε αρκετούς από αυτούς. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο ποσοτικό. Πρέπει επίσης να βρούμε έναν τρόπο να αυξήσουμε την ποιότητα των δεξιοτήτων. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα έχει μεγαλύτερη σχέση με τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Άρα, να μπορεί να προβλέψει τις ε, μελλοντικές ανάγκες και δεξιότητες και να βοηθάει τα όργανα να προσαρμόζονται στον κόσμο που τα περιτριγυρίζει. Πιστεύω ότι τα σχολεία μας, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια μας πρέπει να διασφαλίζουν την απασχολησιμότητα των φοιτητών των. Τον Νοέμβριο πέρυσι άρχισα το πρόγραμμα Rethinking Education, μια νέα στρατηγική που αφορά όλα τα επίπεδα της παιδείας, από την υποχρεωτική παιδεία στο δημοτικό μέχρι την ανώτερη εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση. Η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα συστήματά μας αυτά παιδείας και εκπαίδευση ε, έχουν ελλείψεις. Δεν δίνουν στον κόσμο μόνο τις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, αλλά πρέπει να είναι μορφωμένοι και ως προς τα πολιτιστικά, την έκφραση, τα μέσα, τα ψηφιακά και την πληροφορική, καθώς και τη γνώση ξένων γλωσσών. Σχεδόν 20% όλων των νεαρών Ευρωπαίων δεν, έχουν, δεν γνωρίζουν αρκετή γραφή και ανάγνωση είναι μαζί με τα 73 εκατομμύρια Ευρωπαίων που έχουν μόνο βασικό επίπεδο εκπαίδευσης. Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως είναι η εγκατάλειψη του σχολείου. Ένας σε έξι νέους Ευρωπαίους παρατάει το σχολείο πριν πάρει τις βασικές δεξιότητες. Και έτσι είναι πιο πιθανό να γίνει άνεργος, να μην έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας και άρα αυτό οδηγεί στην ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ο μόνος τρόπος να αντιστραφούν οι τάσεις αυτές είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής παιδείας. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Το ότι τώρα η παιδεία παίζει βασικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη, αναπτυξιακή στρατηγική σημαίνει ότι πρόκειται για σημαντική αλλαγή στον τρόπο σκέψης μας. Σε ένα μήνα, μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Κομισιόν θα παρουσιάσει το σχέδιο συστάσεών της αναχώρα για το 2013 που δίνει έναν οδηγό για τα κράτη-μέλη στις προσπάθειες μεταρρύθμισής τους. Πολλές από τις φετινές συστάσεις θα προβλέπουν βελτιώσεις στην παιδεία. Το 2011, σε αυτές τις συστάσεις αναχώρα, 26 από τις 27 χώρες πήραν συστάσεις επίσης για την παιδεία. Αλλά δεν αρκούν οι μεταρρυθμίσεις. Μια σωστή παιδεία έχει και κάποιο τίμημα. Και αυτό σημαίνει και σωστή χρηματοδότηση όπως ξέρουμε όλοι, η κρίση έχει πλήξει τα δημοσιονομικά μας και πολλές χώρες άρχισαν να μειώνουν τους προϋπολογισμούς τους για την παιδεία. Το 11 και το 12, 9 χώρες μέλη περιέκοψαν τους προϋπολογισμούς της παιδείας κατά πάνω και 11 μεταξύ 1 και 5%. Αυτό είναι μια πραγματική ανησυχία για μας. Η μείωση των επενδύσεων στην παιδεία, της επένδυσης στην παιδεία είναι αντιπαραγωγική. Στην ετήσια, στο ετήσιο έγγραφό μας για την ανάπτυξη το 12 η Κομισιόν ζήτησε από τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην παιδεία. Και πιστεύω ότι η κακή παιδεία είναι ένα κόστος που δεν μπορεί να αποφύγει σήμερα η Ευρώπη. Βέβαια, η κύρια ευθύνη για την ε, μεταρρύθμιση ε, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι των κρατών μελών. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πολλές από τις προσπάθειές του. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα, αν μου επιτρέπετε. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι από τις βασικές ε, ικανότητες που θεωρούνται ζωτικές για τη συμμετοχή στην κοινωνία της γνώσης. Ωστόσο, 48% των Ευρωπαίων ηλικίας 16 έως 74 ετών έχουν χαμηλές δεξιότητες ε, ως προς τα ψηφιακά. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ελλείμματα ε, και αυτή τη στιγμή αρχίζουν να νιώθουν ε, τον αντίκτυπο της γύρασης του πληθυσμού στην αγορά εργασίας μας. Γι' αυτό φέτος θα αρχίσω μια νέα πρωτοβουλία για καλύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Δεύτερον, το Σεπτέμβριο του 2011 κατέθεσα μια ατζέντα για εξυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν στους ε, χαλεπούς αυτούς καιρούς. Μια από τις προτεραιότητες είναι η βελτίωση της ποιότητας ε, διδασκαλίας και εκμάθησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και γι' αυτό συνέστησα ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου που θα κάνει ειδικέ συστάσεις φέτος το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε να εθαρρύνουμε πιο στενές σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων. Τρίτος, τομέας που αξίζει την πλήρη προσοχή μας αυτή τη διαδικασία εξυγχρονισμού. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η συνεισφορά καλής ποιότητας ε, μαθητείας ε, στην απασχόληση των νέων είναι κάτι ευρέως αναγνωρισμένο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κράτη-μέλη με τη χαμηλότερη ενεργία των νέων είναι εκείνα που έχουν συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης ισχυρά, ελκυστικά και με καλή χρηματοδότηση. Είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό όμως χρειάζεται ΣΔΙΤ, χρηματοδότηση από το δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα και κοινή ανάληψη ευθυνών. Αυτό που βλέπουμε στις χώρες με τις μεγαλύτερες επιδόσεις είναι ισχυρή δέσμευση από τις εταιρείε. Γι' αυτό φέτος τον Ιούλιο θα λανσάρουμε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μαθητείας σε συνεργασία πάντα με τον Επίτροπο του κύριο Άντορ. Η νέα συμμαχία θα φέρει κοντά κράτη-μέλη, κοινωνικούς εταίρους, επιχειρήσεις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενεχομένους αυτό που μας ενώνει είναι το κοινό συμφέρον να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση μέσω της μαθητείας. Θα ήθελα τελειώνοντας να σας ε, πω δύο λόγια για το νέο πρόγραμμα Εράσμος για όλους και ε, τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Ο Έρασμος για όλους είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει πολιτικά όσο και οικονομικά στην αναθεώρηση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτασης στην Ευρώπη. Ο Έρασμος για όλους είναι ε, αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής μας κατά της ανεργίας των νέων εφόσον μπορεί να αυξήσει την απασχολησιμότητα των νέων μας ένα μεγάλο τμήμα του προγράμματος θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την κινητικότητα. Εκεί είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Και όχι μόνο για φοιτητέ, αλλά και για μαθητές του σχολείου, διδάσκοντες, ασκουμένους, μαθητευομένους, νέους εργαζομένους και εθελοντές. Κατά κάποιο τρόπο εκδημοκρατίζουμε την πρόσβαση στο πρόγραμμα Εράσμους. Επίσης υποστηρίζουμε φοιτητές που θέλουν να κάνουν μάστερ ε, όλη τη διάρκεια σε άλλη χώρα, ε, δίνοντας μια διευκόλυνση για φοιτητικά δάνεια. Ουσιαστικά το έρασμος για όλους θα φέρει την κινητικότητα σε 4 εκατομμύρια από το 14 μέχρι το 20. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι γνωρίζουμε ότι η κινητικότητα ε, στην εκμάθηση είναι η θύρα που οδηγεί και στην κινητικότητα στην εργασία. Ο κόσμος ε, αποκτά προσόντα που τον βοηθάν να βρει καλύτερες δουλειές. Άρα λοιπόν ένας από τους στόχους και ο υπαριθμόν ένα του Εράσμους για όλους είναι να αυξηθεί το επίπεδο δεξιότητας και να είναι και πιο στοχευμένη για αυτό που χρειάζεται η κοινωνία και οι εταιρείε. Επίση, θα έχουμε πιο καινοτόμε ε, προσεγγίσεις για να μην υπάρχει ανεργία των νέων με ε, εταιρικές σχέσεις διαρθρωμένες μεταξύ εκπαίδευσης και εταιριών. Αυτές είναι οι συμμαχίες για τη γνώση στα πανεπιστήμια και οι ε, ε, κλαδικές συμμαχίες ε, δεξιοτήτων σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό θα είναι δυνατόν να επεκταθεί και σε εθνικό επίπεδο μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Οι διαπραγματεύσεις για το έρασμο για όλους τώρα φτάνουν σε μια αποφασιστική φάση. Εγώ πιστεύω ότι το πνεύμα είναι επικοδομητικό και ελπίζω να επιτύχουμε συμφωνία το συντομότερο. Ωστόσο, θα ήθελα να σας επισημάνω δύο σημαντικά θέματα. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη ευελιξίας. Οι ανάγκες αλλάζουν συνεχώς σήμερα και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα που να μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα στις πολιτικές και οικονομικές πραγματικότητες. Σήμερα, για παράδειγμα, το πρόγραμμά μας δεν μπορεί να ανταποκριθεί με το όσο στένος θα θέλαμε στην ε, ανεργία των νέων. Και αυτό γιατί υπάρχουν εγγενείς αγγυλώσεις Δηλαδή ο προπολογισμό σε μεγάλο βαθμό είναι προκαθορισμένος, εκ των προτέρων προφανώς, ε, για τους διάφορους κλάδους της εκπαίδευση. Γι' αυτό προτείνουμε στο νέο πρόγραμμα Εράσμου για όλους να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία γύρω από ένα σύνολο στόχων που μπορεί να είναι σαφής και συνεκτική. Σε αντίθεση με αυτό, η συγκήτρια προτείνει να αυξηθεί ο αριθμό των στόχων και των δράσεων στο πρόγραμμα και να προκαθοριστούν, να προεγγραφούν 83% των κονδυλίων στους διαφόρους ε, δικαιούχους. Με άλλα λόγια, να διατηρηθεί το status quo. Και αυτό μας φέρνει στο δεύτερο θέμα, το όνομα του προγράμματος. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτό δεν είναι καθόλου επιφανειακό επιπόλαιο, είναι θέμα αρχής μιλούμε για την σύνολη απλούστευση. Αυτό είναι στην καρδιά των προτάσεων, όπου το έρασμο για όλους ε, συνενώνει 7 υφιστάμενα προγράμματα σε ένα σύνολο ε, στρατηγικό και ολοκληρωμένο. Αν συμφωνούμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα πρόγραμμα, ενιαίο, με σαφή πολιτικό στόχο και εστίαση, τότε θα πρέπει να έχουμε και ένα όνομα το οποίο να είναι αξιόπιστο και δημοφιλές και που να συμβολίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πιο αγαπημένα της ιδεώδη. Κατά την άποψή μου, ε, το μόνο όνομα που μπορούμε να δώσουμε είναι έρασμος. Αν θέλουμε να το επεκτείνουμε, να το ανοίξουμε, τότε το έρασμος για όλους στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Είμαι πεπισμένη ότι αν δεν εκμεταλλευτούμε πλήρως το δυναμικό της απλούστευσης και ένα σήμα κατά τεθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αυτό πιο αγαπημένα, τότε θα κάνουμε λάθος. Τέλος, και πραγματικά καταλήγω με αυτό, Πρόεδρε, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στη δράση μας, να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά για την νεολαία μας, τότε θα πρέπει να επενδύσουμε σοβαρά στην εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίω, καλωσορίζουμε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στην πρωτοβουλία ε, που προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την απασχόληση των νέων. Αυτό θα εστιάσει στις περιφέρειες που το χρειάζονται περισσότερο στους νέους και θα βοηθήσει να εφαρμοστεί το σύστημα εγγύσεων για την νεολαία. Αλλά με ένα προπολογισμό 17 δισεκατομμυρίων ευρώ για τον έρασμο για όλους και αύξηση 63% περίπου στην τρέχουσα δαπάνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σαφέστατα τις προτεραιότητές της. Μετά όμως την πρόσφατη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προτείνουμε ένα προπολογισμό 13 δις περίπου, 13,3 για την ακρίβεια. Βεβαίω υπολείπεται ε, των φιλοδοξιών μα, αλλά παραμένει αύξηση του προπολογισμού σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο. Γι' αυτό αξιότιμα μέλη πιστεύω ότι είναι δύσκολε οι διαπραγματεύσει αυτέ, αλλά ελπίζω τελικά να μπορώ να ε, υπολογίζω στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου στον τελικό γύρο των διαπραγματεύσεων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και τώρα ε, περιμένω να ακούσω τα σχόλια και τι ερωτήσει. Ευχαριστώ. Euh, Σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ Επίτροπε, και θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην Αντιπρόεδρό μας, Τσουμπόρα, και στη συνέχεια στην κυρία Μπεναραμπατού. Μπατού. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω την Επίτροπο. Δύο ερωτήσεις θέλω να θέσω. Η πρώτη έχει να κάνει με τον έρασμο για όλους για μένα πέρα από το ζήτημα του ονόματος του προγράμματος αυτού. Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά μπορεί να αλλάξει το πνεύμα του όλου προγράμματος είναι να χορηγεί δάνεια προς φοιτητές. Μάλλον, αυτό έχει, έχει αλλάξει εντελώ τη φύση του προγράμματος. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό είχε μια ιδιαίτερη υποστήριξη στο παρελθόν, αλλά ας μην έχουμε την ψευδέστηση ότι όλοι οι φοιτητέ μπορούν και συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Πολύ συχνά μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν ήδη αρκετά χρήματα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, μπορούν να συμπληρώνουν δηλαδή για να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα αυτό. Ουσιαστικά απευθυνόταν μόνο στους φοιτητές αυτούς οι οποίοι είχαν κάποιου γονεί ευκατάστατους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν τον λόγο να μην δημιουργούμε συνθήκες ανισότητας ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι μπορούν να πάρουν τα δάνεια τα οποία προβλέπονται στα πλαίσια του Εράσμους για όλους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να επιβαρύνει ιδιαίτερα ορισμένους φοιτητέ, οι οποίοι προτού καν αρχίσουν να εργάζονται, πρέπει ήδη να αποπληρώσουν κάποια δάνεια. Νομίζω λοιπόν δεν θα πρέπει να έχουμε αυτή την ανισότητα, δεν θα πρέπει να υποχρεώνουμε τους φοιτητέ να συνάπτουν δάνεια. Διαφορετικά θα πρέπει να προσεγγίσουμε το πρόγραμμα αυτό. Και τώρα κάτι που σχετίζεται πιο ιδιαίτερα με τη χώρα μου, την Πορτογαλία. Όπω θα γνωρίζετε, η Τρόικα ασχολείται ιδιαίτερα με τη χώρα μου αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και ένα από του τομεί που πλήττεται περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι ο τομέα τη εκπαίδευση. Εκεί προβλέπονται περισσότερε περικοπέ στον τομέα δηλαδή της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης και πέρυσι 15.500 άνθρωποι που εργάζονταν στον τομέα της παιδείας απολύθηκαν και 4.500 από αυτούς ήταν καθηγητές, δάσκαλοι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μειωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και καταλαβαίνετε ότι αυτό με τη σειρά του επιβαρύνει ιδιαίτερα τους ίδιους τους εναπομείναντες καθηγητές, καθότι θα αντιστοιχούν πλέον περισσότεροι μαθητές στους καθηγητές αυτούς. Αυξάνεται δηλαδή ο φόρτος εργασίας τους, άλλα σχολεία πάλι έχουν κλείσει. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θέτω είναι ξεκάθαρο κατά την άποψή μου. Σήμερα βλέπουμε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τρόικας και της κυβέρνησης της Πορτογαλίας και προσπαθούν να δούνε πού θα γίνουν περισσότερες περικοπές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τον ε, Ιανουάριο είχε πει ότι θα μπορούσαν περισσότερες χιλιάδες καθηγητές να απολυθούν στην Πορτογαλία. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες περικοπές στον τομέα της παιδείας πρόεδρος. Θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις και θα σας δώσω τη συνέχεια στο λόγο, κυρία Βασιλείου. Νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε πρώτα τους ε, ομιλητές και στη συνέχεια να απαντήσετε εσείς. Αλλά ποιος θέλει να πάρει τώρα το λόγο, θα ήθελα να μου πείτε, για να ξέρω και πόσο χρόνο μιλίας θα έχετε. Η κυρία Μπεναραμπατού πρώτη, ο κύριος Σέρκας, ο κύριος Μπένιον, η κυρία Κοστέλο, θα πάρω και εγώ μετά το λόγο. Και έτσι κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Κυρία Μπεναράμπα, έχετε το λόγο και συνέχεια ο κύριος Σέρκας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένη. Κύριε Επίτροπε, όπως το γνωρίζετε, βρισκόμαστε στα πλαίσια ενός τριμερούς διαλόγου για το πρόγραμμα διαβίου εκπαίδευσης. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα του ονόματος, το όνομα «Έρασμος για όλους» μας κάνει σε εμάς τους πράσινους, αλλά ξέρετε ότι είμαστε μειονότητα. Θεωρούμε ότι είναι καλό το όνομα αυτό για την στιγμή προ τα έξω. Βέβαια, τώρα όσον αφορά τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι το όνομα των δράσεων αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του προγράμματο αυτού. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή δεν διατηρούμε τα επιμέρους ονόματα Λεωνάρτο Κομένιους, αλλά οι δράσεις αυτές είναι πολύ γνωστές από όλους τους δικαιούχους. Εμείς θα θέλαμε να κρατήσουμε στα πλαίσια του Εράσμου για όλους και τις ονομασίες των επιμέρους προγραμμάτων, τα οποία ο κόσμος γνωρίζει, γνωρίζει τους στόχους τους. Το πρώτο σημείο που είναι προβληματικό κατά την άποψή μου είναι ο προπολογισμό για το πρόγραμμα αυτό. Το είπατε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό για την παιδεία, για την εκπαίδευση. Νομίζω ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης, το είπε και η Πορτογαλίδα συνάδελφος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Επιτροπή ε, Πολιτισμού είχε προτείνει 19 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια πρότεινε 17 και τώρα έχουμε φτάσει στα 14 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό δεν αρκεί, πρέπει να το πούμε. Αν θέλουμε πραγματικά να αποτελέσει η εκπαίδευση προτεραιότητα, θα πρέπει να έχουμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Μια χρηματοδότηση που θα ανταποκρίνεται στους στόχους μας. Τώρα, όσον αφορά τις, τα δάνεια αυτά, Είδαμε πω εξελίχθηκε το αντίστοιχο πρόγραμμα στι ΗΠΑ. Πολιτείες. Ελοχεύει ο κίνδυνο να επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τους νέου, οι οποίοι δεν έχουν κάποια εγγυημένη εργασία όταν τελειώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Θα πρέπει να είναι καλά οριοθετημένα, πλαισιωμένα αυτά τα δάνεια. Ξέρω ότι σε πολλέ χώρε υπάρχουν υποτροφίε και αυτό που πιο είναι ότι αν εγκρίνουμε ένα σύστημα δανείων, ενδεχομένω να καταστρέψουμε το εφιστάμενο σύστημα των υποτροφιών, το οποίο βοηθά ιδιαίτερα του φτωχού φοιτητέ να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και ανταυτού τελικά θα έχουμε ένα σύστημα δανείων, το οποίο, όπω σα είπα, θα αποτελέσει ιδιαίτερο άχθο για του φοιτητέ, όταν αυτοί θα αποφυτίσουν από το Πανεπιστήμιο, καθότι θα πρέπει να αρχίσουν να αποπληρώνουν το δάνειο αυτό. Το Συμβούλιο μέχρι στιγμή δεν μα έχει δώσει τι απαραίτητε εγγύσει ότι όντω το πρόγραμμα αυτό σύναψη δανείων είναι σωστά οριοθετημένο και σωστά πλαισιωμένο, να μην επιβαρύνονται ιδιαίτερα οι νέοι όταν τελειώσουν τι σπουδέ του. Κάτι ακόμα το οποίο μα δημιουργεί προβλήματα είναι το ακόλουθο. Έχουμε μία εγγύηση για την νεολαία η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Έχουμε τα διευθυντικά ταμεία και έχουμε και αυτό το σύστημα ανάληψη δράση. Πώ θα καταφέρουμε να διαρθρώσουμε όλο αυτό το σύστημα, πώ θα το χειριστούν τα κράτη-μέλη, σε ποια φάση θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα ή στα πλαίσια των διευθυντικών ταμείων έχουμε την απαραίτητη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό της εκπαίδευσης για τα προγράμματα της ε, νεολαίας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε περισσότερα πράγματα. Πώς θα διαρθρωθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης κατάρτισης. Και μια τελευταία παρατήρηση. Μα έχετε ήδη υποβάλει τρεις ερωτήσεις, λέει η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, σε τρία λεπτά μπορεί κανεί να υποβάλει ακόμα και δέκα ερωτήσει, αλλά θα πρέπει να περιορίσετε κάπω την παρέμβασή σα. Ναι, τελειώνω. Όσον αφορά την ευελιξία, η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να έχουμε το μέγιστο ποσοστό ευελιξία όσον αφορά τι δράσει. Αυτό μα προκαλεί πρόβλημα. Γιατί εμεί θα θέλαμε οι στόχοι να είναι σωστά αναγνωρισμένοι και να μην επιτρέψουμε μια πολύ ευρεία χρηματοδότηση χωρί να γνωρίζουμε ακριβώ ποιε δράσει θα χρηματοδοτηθούν. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρο. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στι τέσσερι βασικέ προποθέσει που έχει θέσει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο έχει θέσει και το ζήτημα τη ευελιξία. Ο Φιλ Μπένιον και συνέχεια η κυρία Κοστέλο. Όχι, μάλλον ο κύριο Θέρκα πρώτα και μετά ο κύριο Μπένιον. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Με έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό οι συνάδελφοι. Μια ερώτηση μόνο για να μην σα φάω και το χρόνο. Το είπε και η συνάδελφο, ε, κυρία Σούμπερ. Η Τρόικα ε, οι μεγάλες ανοησίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Ε, καταστρέφουν ε, τα συστήματα. Εμένα η οικογένειά μου είναι δάσκαλη και στα ισπανικά σχολεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναπληρωτές όταν αρρωσταίνει ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής. Άρρωστος ο καθηγητής ακυρώνεται το μάθημα. Δεν υπάρχει ενισχυτική δασκαλία. δασκαλία. Ε, για ανθρώπους με αναπηρίες, για μετανάστες κτλ. Πέφτει η ποιότητα. Και αυτά είναι οι συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στην Τρόικα, στα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Ποιος είναι το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόνο το Εκοφίνο, ο Επίτροπος κύριος Ρεν, μόνο οι άνθρωποι με τα μαύρα κουστούμια που περιφέρονται στις χώρες μας. Πού είναι οι Επιτροποί, άνδρες και γυναίκες που θα αποτελέσουν το αντίβαρο. Η ε, οι είναι κοινωνικά και κάνουν μια πολιτική για το αύριο, αλλά ξεκινούν τη μακροπρόθεσμη. Συμφωνώ απολύτω με εσά, κυρία Πρόεδρε. Είστε καταπληκτικοί και έχετε και θαυμάσιε ιδέε. Την πολιτική όμω τη χαράζουν άλλοι. Ή μήπω οι υπάλληλοι. Ε, το σώμα των επιτρόπων τι είναι, μόνο για να υπογράφει σε πολιτικέ που καταστρέφουν, κυρία Πρόεδρε, την ποιότητά μα και κυρία Επίτροπε. Και ο κόσμο, ο πιο ευάλωτο υφίσταται αυτέ τι συνέπειε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Merci, Phil Φιλ Μπένιον και κυρία Κοστέλο μετά. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις, κυρίως όσον αφορά τη γενικότερη τοποθέτησή σας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν μιλάτε για τους μακροπρόθεσμους στόχους, ότι όντως θα πρέπει η εκπαίδευση και η κατάρτιση να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και προφανώς τα κράτη-μέλη θα πρέπει να περιορίζουν, να περικόπτουν ε, τον προπολογισμό για την εκπαίδευση ενώ θα πρέπει να κάνουν τελικά αλλού περικοπές, αλλού εφαρμόσουν τα μέτρα λιτότητας. Αυτό λυθεύει απολύτως. Αλλά βέβαια έχω μια πολύ μικρή διευκρίνηση να κάνω προς αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει όχι απλώς να διασώσουμε αλλά και να αυξήσουμε την ποιότητα και την ποσότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα αυξηθεί το κόστος. Ξέρετε ότι η εκπαίδευση έχει να κάνει με τους ανθρώπινους σπόρους, αλλά νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και μια κάποια καινοτομία. Να βελτιώσουμε την ποσότητα και την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας στα πλαίσια των προπολογισμών που ε, έχουμε στη διαθεσή μας. Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τελικά βραχυπρόθεσμες λύσεις στην οικονομική κρίση. Πώς μπορούμε κάπου να δανειστούμε περισσότερα χρήματα, να δημιουργήσουμε μια τεχνητή ζήτηση αλλού, χωρίς τελικά οι άνθρωποι αυτοί να επικεντρώνονται στις διαθροτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Και μία από αυτές τις διαθροτικές αλλαγές είναι μια μεγαλύτερη δέσμευση, μια αύξηση της παρεχόμενη παιδείας και κατάρτιση νομίζω ότι πραγματικά αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τη γενικότερη τοποθέτηση την οποία κάνατε. Και τώρα κάποια επιμέρους ζητήματα όσον αφορά το εράσμο για όλους καθώς επίσης και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Η ομάδα μου, η ομάδα των φιλελευθέρων, σαφώ υποστηρίζει την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. και έχουμε μία μακροχρόνια δέσμευση για το Εράσμος. Και θα θέλαμε και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να ελοποιηθεί σύντομα και θα θέλαμε το πρόγραμμα Εράσμους να εξελιχθεί και να βελτιωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Βλέπουμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολλά ωφέλη και ιδίω ωφέλη όσον αφορά την αποσχολησιμότητα των νέων πτυχιούχων. Ιδίω αυτοί οι οποίοι έχουν πάει σε διάφορε χώρε και δεν έχουν σπουδάσει μόνο στη δική του, έχουν πολλά επιπλέον, πολλές επιπλέον δεξιότητε και όχι μόνο γλωσσικέ δεξιότητε. Και αυτό του βοηθά να βρουν μια θέση εργασία στη συνέχεια. Α μην το ξεχνάμε λοιπόν αυτό. Τώρα, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιε διστάμενε απόψει μεταξύ μου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του προγράμματο, δεν νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είχα να κάνω, δεν υποβάλλω ερωτήσει, αλλά απλώ να κάνω κάποιε παρατηρήσει. Ευχαριστούμε, κυρία Κοστέλο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Νομίζω ότι έχω ήδη καλυφθεί από του προαλήσαντε σε πολλά από τα ζητήματα που ήθελα να θίξω. Ιδίω όσον αφορά την σημασία των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Και χαιρετίζω πραγματικά τη σχετική δέσμευσή σα, κυρία Επίτροπε. Έχω εδώ πέρα μια μοναδική εμπειρία, γιατί έχω εργαστεί σε μια εθνική υπηρεσία για 10 χρόνια, σε μια υπηρεσία προγραμματισμού της Ιρλανδίας και ως προς ε, το πρόγραμμα έρασμος για όλους, πέρα από το όνομα, ως προς την ουσία του κιόλας, θα ήθελα να αφαιρθούμε σε κάποια ζητήματα, κύριε Επίτροπε. Ξεκινήσαμε με το Σόκρατες, έγινε Σόκρατες 2, που ήταν ένα συνολικό πρόγραμμα για πολλά επιμέρους προγράμματα. Στη συνέχεια γίνεται το πρόγραμμα διαβίου μάθησης, το οποίο νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό όνομα από μόνο του, Lifelong Learning Program, το οποίο κάλυπτε τελικά όλη την γάμα, όλη την πορεία εκπαίδευσης ενός ανθρώπου από την αρχή μέχρι το τέλος της ζωής του. Τώρα, το να χρησιμοποιήσουμε μία νέα ονομασία του προγράμματος αφού του συνολικού, δίνοντας το όνομα «Εράσμος για όλους, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί μία σύγχυση. Το «Εράσμος» για πάρα πολλούς ανθρώπους συνδέεται με την ανώτατη εκπαίδευση, το Κομίνιους επίσης είναι ιδιαίτερα γνωστό και ιδιαίτερα δημοφιλές. Πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη γνωρίζουν ποιο είναι το πρόγραμμα Κομίνιους. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά κρίμα αυτή τη στιγμή να χάσουμε αυτέ τι γνωστέ από του Ευρωπαίου πολίτε ονομασίες. η πρόταση που γίνεται αυτή τη στιγμή νομίζω ότι πραγματικά διαβρώνει όλη αυτή την διάσταση, όλη την πτυχή του προγράμματος διαβίου μάθησης για τους ενήλικες. Όταν είχαμε το πρόγραμμα Lifelong Learning, αυτό είχε να κάνει και με την επίσημη και με την άτυπη εκπαίδευση. Ενώ τώρα φοβάμαι ότι με τη νέα ονομασία δημιουργείται τελικά μία σύγχυση. Πολλοί θεωρούν ότι το πρόγραμμα Λεωνάρντο έχει αντικαταστήσει την διαβίου μάθηση για τους ενήλικες. Εν μέρη συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά το πρόγραμμα νεονάρτου ήταν εντελώ διαφορετικό και ξεχωριστό στο παρελθόν. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι δεν τονίζουμε στο υφιστάμενο πρόγραμμα την διάσταση αυτή τη διαβίου μάθηση για του ενήλικε. Μπορούμε να υποστηρίξουμε περισσότερο τη διάσταση αυτή και να καταφέρουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα αυτό ω ξεχωριστό πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Όσον αφορά το πρόγραμμα Εράσμους, σας είπα ποια είναι η δική μου η άποψη όσον αφορά την ευελιξία. Και πραγματικά είναι λυπηρό το ότι δεν καταφέρατε να έρθετε εδώ πέρα νωρίτερα όταν συζητούσαμε στην Επιτροπή μας το ζήτημα της ονομασίας, γιατί και εγώ φοβάμαι ότι το Εράσμους για όλους είναι καλύτερο από ότι το yes, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα. Συμφωνώ Πάντως με όσα είπε η αντιπρόεδρό μας, η ε, κυρία Τσούμπερ, ότι το ζήτημα των δανείων, της σύναψης των δανείων, ιδίω όσον αφορά την πολύ δύσκολη κατάσταση που ζουν πάρα πολλοί νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα προβληματικό σημείο της πρότασης. Θα μπορούσα να κάνω πολλές παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με πολλά πράγματα τα οποία και εσείς θίξατε φοβάμαι ότι δεν αναφέρεστο με σε όλες τις συνέπειε και τι επιπτώσει. Είναι σαφή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εκπαίδευση και η παιδεία. Αυτή την προσέγγιση την έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από την διαδικασία της Λισαβόνας. Και χάρη στα δεδομένα του ΩΣΑ βλέπουμε ότι ήδη πριν από το 2007 το ίμιση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν μειώσει τελικά τον προπολογισμό τους για την εκπαίδευση. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να ασκεί πίεση στα κράτη-μέλη μόνο για το δημόσιο χρέος τους ή για το δημόσιο έλλειμμά τους, θα έπρεπε να ασκεί πίεση και να παρενοχλεί, θα έλεγα, και για το ζήτημα του προπολογισμού που αφιερώνεται στην παιδεία. Μας είπατε ότι η φτωχή παιδεία είναι ένα τίμα το οποίο δεν μπορεί να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα συμφωνώ μαζί σα. Τότε θα πρέπει να μιλήσετε όμω με τον κύριο Όλι Ρεν και να του πείτε ότι κάθε φορά που η Τρόικα πηγαίνει σε ένα κράτο μέλο δεν μπορεί κατά προτεραιότητα να ζητά οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει να λαμβάνουν χώρα και να αφορούν μόνο την το όριο για παράδειγμα, ε, συνταξιοδότησης και να μην αναφέρονται όμω καθόλου στο πόσο θα πρέπει να προωθείται ο τομέας τη εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, επι... να επιτρέπεται να επηρεάζει τελικά τον προπολογισμό της εκπαίδευσης για να διορθωθούν τα δεδομένα για το δημόσιο έλλειμμα. Συμφωνούμε, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι είναι μια προστιθέμενη αξία με την οποία θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, όπως την ανταγωνιστικότητα, την, παγκοσμιο... παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να επενδύουν περισσότερο στην εκπαίδευση, στα συστήματα παιδεία. Διαφορετικά ουσιαστικά οι όλε αυτέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτελέσουν μπούμεραν για τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τι ψηφιακέ ε, δεξιότητε. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η χώρα της Βαλτική, Πάντω θα το γνωρίζετε κι εσείς, ότι ετέθη το ζήτημα της εκπαίδευσης όσον αφορά τις ε, ψηφιακές δεξιότητες και αυτό αποτελεί τμήμα ήδη της δευτερο, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή οι άνθρωποι, τα παιδιά στη χώρα αυτή μαθαίνουν μαθηματικά, μια δεύτερη ξένη γλώσσα και μαθαίνουν και πληροφορική, μια γλώσσα πληροφορικής. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν καλό να είχαμε μια σχετική κατευθυντήρια γραμμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναβερθήκατε επίσης πολύ στην μαθητεία. Και ξέρετε ότι και εμείς εδώ σε αυτή την Επιτροπή θαυμάζουμε πραγματικά τις χώρες αυτές, όπως είναι η Αυστρία, και η Γερμανία, οι οποίες διαπρέπουν στο ζήτημα της μαθητείας. Αυτό όμω που είδαμε είναι ότι στις χώρες αυτές είναι παραδειγματική μαθητεία, γιατί τελικά βασίζεται και στο ζήτημα της ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου και ότι υπάρχει μια καλή διάρθρωση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τον εκπαιδευτικό τομέα, ο οποίος όμως δεν είναι θεωρητικός, αλλά είναι και ποιοτικός, είναι ουσιαστικός ξέρετε ότι δεν μιλάμε απλώς έτσι για τον κοινωνικό διάλογο. Ο κοινωνικός διάλογος δεν μπορεί να δρεωθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν πραγματικά θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το τομέα. Τέλος, αναφερθήκατε στο ζήτημα της κινητικότητας. Προφανώ και εμεί γνωρίζουμε ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην όλη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωση, και ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των βασικών ελευθεριών τη συνθήκης της Ρώμης. Στα πλαίσια όμως υφιστάμενη οικονομικής κρίσης, η έννοια της κινητικότητας θα πρέπει να αναθεωρηθεί υπό το φως της κρίσης αυτής και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι εννοούμε όταν λέμε κινητικότητα. Το πρόγραμμα Εράσμους είναι ένα πρόγραμμα, αν θέλετε, της περίοδος των παχαίων αγελάδων. Σε περίοδο κρίσης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί, αλλά θα πρέπει να δούμε παράλληλα και ποια είναι η πραγματική κινητικότητα τελικά των νέων. Σαφώς η κινητικότητα η θελούσε κινητικότητα έχει προωθήσει πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξέρετε ότι υπάρχει και μία κινητικότητα επιβεβλημένη πολλές φορές, ακούσια, η οποία είναι σαφώς αρνητική. Και ξέρετε ότι πολλές φορές η κινητικότητα αυτή η υποχρεωτική τελικά, ξεκινάει από τις χώρες εκείνες οι οποίες έχουν προβλήματα δημοσιονομικά, τα οποία επιδεινώνται περισσότερο από ορισμένε πολιτικές της Τρόικας, όπου ορισμένοι πολίτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες αυτές, να εργαστούν σε μία άλλη χώρα και επιστρέφουν στη χώρα τους μόνο για να πάρουν τη σύνταξή τους, μάλλον στην ηλικία της συνταξιδότητας πια. Δεν μπορούμε να προωθούμε εμεί μία τέτοιου είδους κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορά που μιλάμε για κινητικότητα θα πρέπει η κινητικότητα αυτή να είναι θετική και να αποτελεί τελικά πλεονέκτημα για τους νέους Ευρωπαίους. Βλέπετε λοιπόν ότι οι συζητήσει που γίνονται στην Επιτροπή μα είναι πάντα ιδιαίτερα ενθουσιώδει και έντονε. Ελπίζω να μην έχετε μετανιώσει που είστε εδώ και περιμένουμε τώρα να ακούσουμε τι απαντήσει σα. Let me start with... Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από ένα σημείο που ανέφεραν πολλοί η εγγυημένη διευκόλυνση για δάνεια για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιτρέψτε μου να πω ότι ευθύ εξ αρχής αυτό δεν επινοήθηκε ως ένας τρόπος να αποφευθούν οι ε, υποτροφίες. Οι υποτροφίες θα παραμείνουν βασικός μας στόχος. Και μακάρι να είχαμε τον απαραίτητο προϋπολογισμό για να δώσουμε υποτροφίες και για μεταπτυχιακούς ε, στο εξωτερικό. Αυτό θα ήταν ιδεώδης ε, κατάσταση. Αλλά εμείς ανταποκρινόμαστε τώρα σε μια ανάγκη. Έτσι, αντιδρούμε σε μια ανάγκη, διότι είπα και στην εισαγωγή μου ότι γνωρίζουμε ότι στο μέλλον το 35% των θέσεων εργασίας θα απαιτούν υψηλά προσόντα. Δηλαδή μεταπτυχιακά. Και όπως όλοι γνωρίζουμε. Σήμερα ποιος παίρνει δάνειο για μεταπτυχιακό. Εκείνοι που μπορούν να πάρουν δάνειο και να δώσουν και ε, εμπράγματες εγγυήσεις των γονέων ας πούμε και έτσι παίρνουν τα δάνεια. Μα γι' αυτό επειδή θέλουμε εμείς να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη διευκόλυνση εγγύησης των δανείων γιατί ελπίζουμε έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα στους λιγότερο ευνοημένους να ταξιδεύουν και να κάνουν μεταπτυχιακά χωρίς να έχουν την υποχρέωση να ζητήσουν από τους γονείς τους αυτή την χρηματική ασφάλεια. Και επίσης, εξασφαλίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλή η όρη για τους φοιτητές. Πρώτον, δεν θα καταχρεωθούν οι άνθρωποι. Λέμε το πολύ 12.000 ευρώ για ένα έτος ε, σπουδώνει 18.000 για μια διετία, όταν είναι το μάστερ διετές. Και αυτό μπορεί να μπει και σε ένα παράρτημα. Δεν θα απαιτούνται επιπλέον εγγυήσει σε πράγματες, είτε από τους γονείς είτε από τους ίδιους. Τρίτον, πάρα πολύ ευνοϊκό επιτόκιο και μια περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή και σε περίπτωση ε, που χρειαστεί να υπάρχουν και δυνατότητες διακοπής αναστολής και ε, κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής με δόσεις. Εντάξει, γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα γι' αυτό και ε, σε μεγάλες λεπτομέρειες κυκλοφορεί μια ιδέα ότι μπορεί να χρειαστεί μια δοκιμαστική περίοδος για να δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα και το 2017 να κάνουμε μια αξιολόγηση και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσει μας και να το συνεχίσουμε να το διακόψουμε. Πάντως, πρέπει να πω το εξή. Ακόμα και αν υπάρξει αυτή η δοκιμαστική περίοδος, χρειάζεται και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό για την περίοδο αυτή για να δούμε αν ε, πιάνει ή όχι, αν έχει κάποιο αντίκτυπο. Έτσι, αυτή είναι η εξήγηση που δίνω για τα δάνεια οι περικοπές στον προπολογισμό για την εκπαίδευση. Νομίζω το είπα ξεκάθαρα. Στην ετήσια ε, ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρακολουθεί την ανάπτυξη λέμε ξεκάθαρα ότι τα κράτη θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση ακόμα και όταν εξηγιαίνουν τα δημόσια οικονομικά τους. Δεν μπορούμε βέβαια να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να προβούν σε κάποιες ενέργειες. Ακόμα και στις ειδικέ συστάσεις που κάνουμε ένα χώρα, σε πολλές περιπτώσεις, κάνουμε μια σύσταση που λέγει ότι προσοχή, κάνετε περικοπές στην παιδεία και αυτό θα έχει αρνητικά αποτελέσματα τα οποία θα έρθετε να διαπιστώσετε μετά από λίγα χρόνια. Αλλά είμαστε όλοι ρεαλιστές. Οι εθνικοί πολιτικοί δεν θέλουν άμεσα αποτελέσματα, βλέπουν. Και η παιδεία δεν είναι ένας κλάδος που μπορούν να δουν άμεσο αποτέλεσμα. Γι' αυτό πέφτει εκεί ψαλίδι. Μα γι' αυτό πρέπει να το εξαιρέσετε από το, το σύμφωνο σταθερότητας, λέει η Πρόεδρος. Να μην θεωρούνται δαπάνες οι επενδύσεις στην παιδεία. Ναι. Ε, κάτι ακόμα. <laughs> Επένδυση στην παιδεία δεν σημαίνει αναγκαστικά αύξηση των δαπανών η σοφή επένδυση είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Διότι σε πολλά κρατημέλη, στην πατρίδα μου για παράδειγμα, έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στην εκπαίδευση. Αλλά δεν είμαστε πολύ αποτελεσματικοί διότι δεν επενδύαμε συνετά και με... Σοφία, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητές μας και να επενδύσουμε ε, με πιο μεγάλη σύνεση και ε, σκόπιμα. Ξέρω ότι αυτό συμβαίνει σε πολλά Ε, συμφωνώ πολύτως με αυτό που είπατε σχετικά με τις ποσοτικές αυξήσεις στην παιδεία. Δεν αρκεί η ποιότητα, είναι το πιο σημαντικό. Διότι σήμερα τι παρατηρούμε σε πολλές χώρες το φαινόμενο αυξάνεται η ανεργία μεταξύ των πτυχιούχων. Αυτό δεν είναι ικανοποιητικό, διότι τι νόημα έχει να βγάζεις πτυχιούχους για να είναι άνεργοι. Γι' αυτό πραγματικά θα πρέπει να βάλουμε την έμφαση στην ποιοτική εκπαίδευση. Γι' αυτό ε, και διόρισα την ομάδα υψηλού επίπεδου για εξυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γι' αυτό βάζω και μεγάλη έμφαση ε, στη βαθμολογία των πανεπιστημίων για το ranking αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται ως κριτήριο και η ποιότητα της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας που παρέχεται. Αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμα από την ποσότητα. Now, um, about the name. Για το όνομα του προγράμματος τώρα και τη δομή του νέου προγράμματος. Νομίζω σας εξήγησα γιατί επέλεξα το όνομα Έρασμος για όλους. Διότι από τις μελέτες μας τι βλέπω. Το Κομένιος, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα σχολεία. Το Γκρούντβιχ, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι χιλιάδες που συμμετέχουν, δικαιούχοι. Λεωνάρδο, το αυτό, για τους μαθητευομένους και τους ασκουμένους. Αλλά το έρασμος το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει ουδής ε, είτε Ευρωπαίος είτε εκτός Ευρώπης, άνδρα ή γυναίκα, που να μην έχει ακούσει και να μην εκτιμά και το όνομα. Ένα όνομα έπρεπε να επιλέξω για λόγους απλούστευσης. Αλλά σε ό,τι αφορά τώρα τα υποπρογράμματα, τα επιμέρους, ε, κατανοώ ότι το καθένα, πώς να το πω, καθένας ανησυχεί για το πρόγραμμά του. Είναι συντηρητική, λέει η Πρόεδρος. Εντάξει, μπορεί να είναι και συντηρητική, αλλά είναι δεμένη με τα προγράμματα, αλλά το πρόγραμμα τώρα είναι πολύ διαφορετικό στη δομή του. Έχει εγκάρσια δομή πλέον, όχι κάθετη. Σε κλάδους, κολόνες, ξέρω εγώ, πυλώνες. Έχουμε οριζόντια τώρα κατανομή με τρεις βασικές δράσεις. Κινητικότητα, εταιρικές σχέσεις και υποστηρικτικές πολιτικές. Είτε είσαι μαθητής, είτε είσαι φοιτητής, είτε είσαι εκπαιδευτικός ή εκπαιδευόμενος, θα επιλέξεις ένα από τα τρία. Έτσι το έχουμε τώρα διαρθρώσει. Εάν επιπλέον τώρα διατηρήσουμε και τα υποπρογράμματα, θα γίνει σταυρόλεξο. <laughs> Πολύ πιο περίπλοκο. Άμα έχουμε και οριζόντια και κάθετα. Και έτσι δεν ανταποκρινόμαστε στη βασική μας ευθύνη. Που κατά τα άλλα ξέρετε ήταν και αίτημα του Κοινοβουλίου. Απλούστευση, απλούστευση, απλούστευση. Ε, τι θα πει απλούστευση. Να είναι πιο απλή ε, η λειτουργία παντού. Και υπέρ των δικαιούχων και υπέρ των διαχειριστών και υπέρ όλων των ενδιαφερομένων. Τώρα για τις μαθητείες. Μίλησα πολύ για αυτό το θέμα γιατί πιστεύω <clears throat> ότι έχουμε μια ευθύνη να, την να τις προωθήσουμε. Βλέπουμε από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης πόσο σημαντικές είναι και πόσο απαραίτητο είναι να διατηρήσουν τις θέσεις του οι μαθητευόμενοι. Γι' αυτό έχουμε κάνει μνημόνιο με τις χώρες αυτές και τις νότιες χώρες και γι' αυτό ζητούμε αυτήν την συμμαχία για τις μαθητείες που λέμε για να συνδυάσουμε όλους τους παράγοντες, την Κομισιό, τα κράτη-μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, πολύ σημαντικό, για συνεργασία και για να υπάρξουν περισσότερες μαθητείες και μάλιστα ποιοτικέ. Αυτό θέλουμε. Τέλος για την κινητικότητα. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά που είπατε, γιατί και για μας η κινητικότητα σημαίνει να δώσει κανείς την ευκαιρία στον κόσμο να πάρει αυτές τις οριζόντιες δεξιότητες που χρειάζεται για να βρει δουλειά. Γιατί ακόμα και αν έχει κανείς μια εξαιρετική μόρφωση πανεπιστημιακή, δεν έχει αυτές τις δεξιότητες που θα μπορέσει να πάρει από την κινητικότητα. Γι' αυτό θέλουμε να αυξηθεί η κινητικότητα υπό τον έρασμο. Δεν το κάνω για να ενθαρρύνω brain drain, δηλαδή διαρροή εγκεφάλων, αλλά γιατί αν ένας νέος είναι άνεργος και μπορεί να βρει δουλειά σε γειτονική χώρα, γιατί να μην το κάνει για μερικά χρόνια τουλάχιστον. Δεν είναι όμως αυτός σκοπός. Είναι μια λύση στην περίπτωση που θα χρειαστεί. Ο στόχος μας είναι η απόκτηση των δεξιοτήτων που μπορεί να πάρουν από την κινητικότητα. Thank you very much. I think uh, it was a first exchange. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων από τον διορισμό σας. Ελπίζω όμως να μην είναι και η τελευταία. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων γιατί ουσιαστικά γεφυρώνονται και αυτά τα ζητήματα ανάμεσα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις θέσεις εργασίας. Επομένω, η δική σας συμβολή είναι πολύ σημαντική και για τη δική μας την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή έκβαση στον τριμερή διάλογο.